Λήξε η συνεδρίασή των. Έχουμε εγκρίνει την ημερήσια διάταξη για τις 18-19 Απριλίου. Αναθεωρημένη πρόταση επίσης και η γραμματεία θα εξετάσει το ενδεχόμενο να περιλάβει μια, έναν αριθμό μάλλον ε, αναφορών για την προστασία των ζεών και ιδίως για την κοπή των ουρών των χείρων. Ε, η ομάδα EFTD έχει ζητήσει για τις 2 Ιουνίου θα υποβληθεί μάλλον αίτημα των πράσινων για την 20η και 21η έκτου και επίσης άλλη αίτηση των πράσινων πάλι για θέμα για την δεύτερη σύνοδο του Ιουνίου. Και Έχουμε και την ετήσια έκθεση για το 2015 και την έκθεση της διαμεσολαβήτριας, δηλαδή της συνηγόρου του πολίτου, που θα αναλάβει ο ECR στο πρόσωπο του κ. Μαριά. Και τώρα, για επιλογές για την βελτίωση της πρόσβασης στα φάρμακα έχει εγκριθεί και οι σχετικές συστάσεις έγιναν δεκτές με εξαίρεση μιας αναφοράς όπου οι συντονιστές συμφώνησαν σε συμβαστική πρόταση δική μου, δηλαδή αυτή να διαβιβαστεί προς ενημέρωση στην Επιτροπή Εξωτερικών. Συμφώνησαν να συνεχίσουν με την πρακτική ο δε κ. Κρίστιαν Κνούτσεν, Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Προεδρίας, ήταν παρόν για να συζητήσει τα περί λίστας 3 επίσης για την ελεύθερη διακίνηση και για τις συμβάσεις περιορισμένου χρόνου. Απόφαση θα ληφθεί μετά την ακρόαση σχετικά με κολλήματα δηλαδή για τη διακίνηση των πολιτών στην ενιαία αγορά που θα οργανωθεί η ακρόαση αυτή δηλαδή το φθινόπωρο του 2016. Τα αιτήματα αυτά θα συζητηθούν λοιπόν μετά από την οργάνωση της ακρόασης. Το υπαριθμόν 6, ομάδα εργασίας για την προστασία των παιδιών. Η κυρία Ελεονόρα Εύη αναφέρθηκε στις διαδικασίες της ομάδας εργασίας, την περιοδικότητα των συνεδριάσεών της και κατέστη σαφές ότι τελικώς θα συντάξουν έκθεση στο τέλος των εργασιών τους. Το Λαϊκό Κόμμα ζητεί να κλείσουν ορισμένες αναφορές. Κοιτάξτε, υπάρχει κατάλογος αναφορών που ε, συστήνει και η γραμματεία να κλείσουν και να μεταφερθούν όλες στη λίστα Β. Όλες οι υπόλοιπες αναφορές να ε, αξιολογηθούν σύμφωνα με τις συστάσεις της γραμματείας. Έγινε και ερώτηση από το Λαϊκό Κόμμα σχετικά με την 570 του 13 αναφορά. Εκεί θα αποσταλεί επιστολή στον αρμόδιο επίτροπο για περαιτέρω διερεύνηση και για ε, διερεύνηση Τη ενδεχόμενη παραπέρα πορείας. Η ομάδα των πράσινων τώρα υπέβαλε αίτημα για το follow-up για, την, για το ψήφισμα για, τις, για τους ανθρώπινους πόρους και για τι περιόδου τις περιόδους συνεδριάσεων. Θα στείλουμε επιστολή και με αντίγραφο στον Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης IPOL, που θα συντάξει η Πρόεδρος, εγώ δηλαδή, για το δίκτυο το, της Επιτροπής Αναφορών, Petty Network, θα τα ξανασυζητήσουμε στις 22 Μαρτίου. Μέχρι τότε μπορούν να κατατεθούν προτάσεις από τα μέλη. Οι δε αποφάσεις θα ληφθούν στην ε, συνεδρίαση του Απριλίου. Για το πρόγραμμα εργασιών του ελεγκτικού συνεδρίου προβλέπεται προθεσμία για την υποβολή γραπτών σχολείων μέχρι τις 22 Τρίτου. Ευχαρίστως λοιπόν εκεί να υποβάλλετε προτάσεις. Αυτά αποφάσισαν οι συντονιστές στη συνεδρίασή τους. Και νομίζω λοιπόν ότι είμαστε τώρα πια έτοιμες να προχωρήσουμε στο πρώτο θέμα της σημερινής ημερησίας διατάξεως που προβλέπει ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε φέρει τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας. Όλοι και όλες, ωραία. Πρόταση ψηφίσματος, ίσως μάλιστα να βγάλω και εγώ την κάρτα μου, έτσι είναι. Κοιτάξτε, όπως είπα, αν έχετε όλες τις, ε, την ε, κάρτα ψηφοφορίας, πρόκειται για την προστασία των συμφερόντων του παιδιού σε διασυνοριακές υποθέσεις. Πρώτα, αιτιολογική σκέψη α σε δύο τμήματα. Ψήφι υπέρ του πρώτου τμήματος. Εγκρίνεται. Τμήμα δεύτερο, υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αυτό. Τώρα, αιτιολογική σκέψη δέλτα. Α, μόνο ένα, ε, τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 3 τώρα. Προβλέπεται, προβλέπονται δύο τμήματα μάλλον. Πρώτο τμήμα, υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ελπίζω ότι λειτουργεί. Α, φαίνεται πως δεν λειτουργεί το μηχάνημα. Ωραία. Τώρα. Τέλος της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά Α, ήταν ήδη το δεύτερο τμήμα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Όπως αντιλαμβάνεστε μόλις βγαίνω από τους συντονιστές και έχω λίγο ζαλιστεί. Παράγραφος 11, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία για την επαλήθευση. Τέλος. Απορρίπτεται. Με μια ψηφοδιαφορά. Ασύνηθες. Παράγραφος 9. Σε τρία τμήματα. Πρώτο, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται βεβαίως, σαφώς. Ε, τμήμα τρίτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται και αυτό. Παράγραφος 10. Υπέρ. Α, πρώτο τμήμα, ε. πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Επαλήθευση έχει καλώς. Αρχίζει. Πέρας. Έγκρινεται λοιπόν. Δεύτερο τμήμα. Όχι. Όχι, με συγχωρείτε. Παράγραφος 23, πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αρχίζει. Τέλος. Απερίφθη. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έχει καλώς. Αυτή λοιπόν ήταν η ψηφοφορία. Μην ξεχάσετε τις κάρτες σας μέσα στην σχισμή. Και ακολουθεί η αναφορά που έχουμε σήμερα, η 0336 του 15 για κρατικές ενισχύσεις που έχουν ληφθεί από την εταιρεία ASP. Τζάνι Σερβόνη, αναφερόμενος, είναι εδώ κοντά μας και τα μέλη που επιθυμούν να εξέλθουν από την αίθουσα. Έχει καλό, σας περιμένουμε λίγα δευτερόλεπτα μέχρι ότου το πράξουν. Παρακαλούνται τα μέλη που αποχωρούν τις αιθούσεις να το πράξουν ησύχω για να δώσουμε το λόγο στον αναφερόμενο. Κύριε Σερβόνε, έρχεται το μικρόφωνο για πέντε λεπτά. Θα βάλουμε και το χρονόμετρο σήμερα. Βεβαίως υπάρχει και η μετάφραση. Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το θέμα της γλώσσας. Πέντε λεπτά. Ναι, ναι. Καλή σας μέρα εξ ονόματος των εργαζομένων στους αερολιμένες ε, ε, της Μαλπένσα ε, και του Μιλάνου θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί δεχτήκατε και θεωρήσατε παραδεκτή αυτήν την αναφορά που εκπροσωπεί και αφορά εκατοντάδες εργαζομένους. Ήδη το Δεκέμβριο του 2012 αποφασίστηκε ότι η Ιταλία θα έπρεπε να επιστρέψει τις ε, επιδοτήσεις ε, που παράνομα είχαν δοθεί στην Sea Handling. Ε, όλο αυτό το θέμα όμως θεωρήθηκε ότι, θεώρησε ότι δεν θα πρέπει να προωθηθούν τα θέματα γιατί μονάχα καλό θα μπορούσε να προκύψει για τους εργαζόμενους. Όμως οι εργαζόμενοι αναγκάστηκαν να κάνουν μεγάλες οικονομικές, κοινωνικές και, και οικογενειακές θυσίες ε, και ε, οπωσδήποτε αυτοί οι οποίοι κέρδισαν είναι ε, οι εκπρόσωποι της e-handling καθώς επίσης οι περιφερειακές τοπικές αρχές αλλά ακόμα και η ίδια η Ιταλική κυβέρνηση η οποία καθόλου δεν κινήθηκε. Όλοι αυτοί γνώριζαν ότι ήδη το 2006 είχε ξεκινήσει μια διαδικασία επιπαραβάση από την Ευρωπαϊκή Ένωση απέναντι στην εταιρεία Sea Handling. Κανείς όμως δεν ανέλαβε την παραμικρή ε, πρωτοβουλία έτσι ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση της ε, εταιρεία αυτής. Μάλιστα, οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των, της ε, εταιρεία έλαβαν σημαντικές θέσεις στην κοινωνία, λες και δεν συνέβη τίποτα, ενώ ξέρουμε ότι δεν έκαναν τίποτα έτσι ώστε να αποφύγουν την πτώχευση. Λαμβάνοντας υπόψη την υπόθεση c Handling, αυτή αρχίζει να γίνεται γνωστή το 2012 όταν η Ευρωπαϊκή ε, ε, Επιτροπή επέβαλε ένα πρόστιμο. Αυτό από την στιγμή που επευλήθη το πρόστιμα ε, ξεκίνησαν διάφορες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και της ε, Ιταλικής κυβέρνησης ανάμεσα στην ΣΥΑ και την Ιταλική κυβέρνηση ανάμεσα στην Ιταλική και την Ευρωπαϊκή Ένωση ανάμεσα στην Ιταλική κυβέρνηση και τα συνδικάτα ανάμεσα στην περιφέρεια και την ΕΣΕ. Ωστόσο και σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου του Λουξεμβούργου αλλά και του Τάρτου Μιλά ε, δεν ε, ε, μπόρεσαν οι εργαζόμενοι να βρουν το δίκιο τους. Αντιθέτως δε διελήθη η παλαιά εταιρεία, δημιουργήθηκε δε μια νέα με, το, με την ονομασία Airport Handling. Θα ήθελα να σας δώσω εδώ κάποια σημαντικά στοιχεία. Η Sea Handling είχε 2.314 εργαζόμενους τη στιγμή ε, της πάυσης των δραστηριοτήτων της. Όταν, ξεκίνησαν, ε, όταν ξεκίνησε τις δραστηριότητες της ε, η νέα εταιρεία, οι εργαζόμενοι ήταν 1.900 και τώρα έχουν γίνει 1.700 άτομα, ενώ ταυτόχρονα έχει αυξηθεί κατά πολύ η κυκλοφορία στα λόγω αεροδρόμια. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι έχουν ιδιαίτερα ιδιαίτερο φόρτο εργασίας. Ειδικά δε οι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι στα γκισέ του τσεκίν, καθώς επίσης και στις ε, αποσκευές, ε, αυτοί υποφέρουν περισσότερο από τους άλλους. Πρέπει να πούμε ότι οι νέοι εργαζόμενοι της νέας ε, εταιρείας δεν έχουν ούτε κάλυψη των κοινωνικών τους, των κοινωνικών τους δικαιωμάτων και υπάρχουν και επίσης για άλλα προβλήματα όπως ας πούμε η μη τήρηση ε, των αρχών ασφαλείας. Για να μην αναφέρω το γεγονός ότι οι νέοι εργαζόμενοι ε, δεν ε, λαμβάνουν την απαραίτητη κατάρτιση και δεν έχουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Όλα αυτά τα έχουν καταγράψει και τα έχουν καταδείξει οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ωστόσο δεν υπάρχει καμία διαφάνεια όσον αφορά τι πληροφορίες τις οποίες έχουν πρόσβαση τα ε, συνδυα Είναι αυτό μονάχα. Πρέπει να πούμε ότι ε, έγινε ψηφοφορία ε, ε, μεταξύ των εργαζομένων οι οποίοι με κανένα τρόπο δεν εδέχοντο τις προτάσεις της εργοδοσίας. Ωστόσο το αποτέλεσμα αυτού του δημοψηφίσματος αυτής της ψηφοφορίας απλώς αγνοήθηκε. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι βρίσκονται στο κέντρο αυτής της παράλογης κατάστασης ζητούν από σας να κατανοήσετε ότι εδώ και δύο δύο χρόνια περιμένουμε, είμαστε σε κατάσταση αναμονής. Μετά από την απόφαση του Λουξεμβούργου δεν έχει κινηθεί τίποτα. Περιμένω λοιπόν απάντηση στις ερωτήσεις τις οποίες ε, είχαμε ήδη στείλει στην Επιτροπή σας, αλλά ε, επίσης και κυρίως θα έλεγα να αναλάβετε δράση έτσι ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια λύση στο πρόβλημά μας. Αναρωτιέμαι τι η Ευρώπη είναι αυτή η οποία δεν μπορεί να παρέμβει σε μια κατάσταση όπου εκατοντάδες εργαζόμενοι απολύουν ο μια Ευρώπη η οποία δεν μπορεί να μελετήσει κατά πόσον τα χρήματα που έχει δώσει έχουν χρησιμοποιηθεί υπέρ των εργαζομένων και υπέρ της διατήρησης των θέσεων εργασίας. Θα δώσω τώρα το λόγο, λέει η Πρόεδρος, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μπερνάρτ Φόντλαντ. <clears throat> Ähm, ähm, ähm, Είναι αληθές ότι έχει ξεκινήσει μια επίσημη διαδικασία εξετάσεως ήδη από το 2012 σχετικά με παράνομες και μη νόμιμες ε, κρατικές επιχορηγήσεις, κρατικές επιδοτήσεις μάλλον προς την ε, Sea Handling. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, η ΔΕ Κομισιόν ζήτησε από την Ιταλική Δημοκρατία να απαιτήσει επιστροφή των ενισχύσεων από την EC Handling. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έχει ρευστοποιηθεί, άρα έχει πτωχεύσει η EC Handling και μετά ξεκινά ή επιδιώκει νέα διαδικασία για να εξετάσει αν η Airport Handling απολαμβάνει πλέον τις επιδοτήσεις αυτές. Δηλαδή αν μεταφέρθηκαν αυτές σε αυτήν. Η διαδικασία αυτή επίσης έχει ολοκληρωθεί και τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται απόφαση επί της ουσίας. Απόφαση η οποία στα πλαίσια της οποίας δηλαδή θα αποφανθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν η ενίσχυση αυτή δόθηκε παραπέρα στην airport handling ή όχι. Όποια και αν είναι η τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αυτό εγώ δεν μπορώ να το προκαταλάβω. Όμως, εξακολουθεί να ισχύει ότι η απόφαση για ανάκτηση εξακολουθεί να ισχύει. Εξακολουθεί να ισχύει δηλαδή ότι η CR Handling καλείται να αποδώσει τις μη νομίμως καταβληθήσεις ενισχύσεις. Γνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια ότι τώρα έχει αναλάβει η Airport Handling και η Sea Handling έχει πτωχεύσει. Σε ό,τι αφορά τώρα τις ενδεχόμενες κοινωνικές επιπτώσεις, η έρευνα που διεξάγεται δεν παρεμβαίνει στις αρμοδιότητες των αρχών που εξετάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού, αν δηλαδή υπάρχει ενδεχομένω παράνομο πλεονέκτημα ανταγωνισμού υπέρ της airport handling. Η προσπάθειά μας είναι να ολοκληρώσουμε ταχύτερον δυνατό την διαδικασία και να εγκρίνουμε σχετική απόφαση όσο δυνατόν ταχύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η πρόεδρος Βίκστρομ. Έχουν δυνατότητα τώρα να λάβουν οι συνάδελφοι τον λόγο. Πέτερ Γιάρ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύσκολο πρόβλημα, πράγματι. Αφενός, όπως εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μπορεί να πει κανείς πού βρίσκεται εν τέλει το πρόβλημα. Εάν κάποιος έχει λάβει αχρεωστήτως ή τέλος πάντων αδικαιολογήτως κάποιες επιδοτήσεις, οφείλει να τις επιστρέψει. Βέβαια, αυτά έχουν κοινωνικές επιπτώσεις και γι' αυτό στρέφονται οι αναφερόμενοι προς εμάς. δεν έλαβαν τις επιδοτήσεις αυτές οι ίδιοι απασχολούμενοι, αλλά η εταιρεία. Και γι' αυτό ζητεί ο αναφερόμενος να ληφθούν υπόψη αυτά. Η ΔΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζητεί, όπως μας εξήγησε. Εγώ νομίζω να παρακαλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη τις επιπτώσεις αυτές. στο νομοθετικό προστάσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και, άλλα, και άλλοι τρόποι για να μειωθούν ε, οι αρνητικές συνέπειες. Γι' αυτό ζητώ να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά και να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι γνωρίζει ότι πρόκειται για παρανόμως ε, εκχωρηθήσεις ενισχύσεις, αλλά να δει πώς μπορεί να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ Πέτερ. Βάλει, πρώτη φορά σας βλέπω. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μελέτησα λίγο το θέμα, αλλά δεν είναι σαφές κάτι. Δηλαδή, εσείς ε, αναφέρεστε ε, στη, στα θέματα που είναι, ας πούμε, ε, το δίκαιο του ανταγωνισμού και το κατά πόσον οι, οι ενισχύσεις αυτές ήταν σωστές ενισχύσεις ή όχι. Αναφέρομαστε όμως στην SEA Handling τώρα η πρώτη εταιρεία ήταν αυτή η οποία το 2000, από το 2002 μέχρι το 2010 ε, είχε ένα παθητικό της τάξης των 380 εκατομμυρίων ευρώ. Από τις πληροφορίες τις οποίες έχουμε αυτό ακριβώς οφείλεται στην κακή διαχείριση της ε, εταιρεία, κακή διαχείριση επίσης ε, την οποία, στην οποία συνέβαλαν και πολιτικές, πολιτικά κόμματα τα οποία οδήγησαν στην ουσία σε αυτή την κατάσταση γιατί είχαν μια ιδιαίτερα ε, χαλαρή στάση απέναντι στους ε, ε, διαχειριστές, τους επικεφαλείς της εταιρείας αυτής. Δεν γινόταν δηλαδή κανενα έλεγχος στην εταιρεία αυτή. Και τώρα έρχεται μια απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία κυρώνει οπωσδήποτε τους εργαζόμενους αλλά με κανένα τρόπο δεν, υφίσταται, δεν υφίστανται καμία κύρωση η πραγματική υπεύθυνοι ε, για αυτή την κατάσταση. Στην ουσία δηλαδή ε, δίνεται, ε, παίρνετε μία απόφαση εσφαλμένη γιατί θα έπρεπε να πάρετε μία απόφαση η οποία να βοηθάει τους εργαζόμενους και να επιβάλλει κυρώσεις στους υπεύθυνους γιατί εσείς βρίσκεστε σε μία κατάσταση όπου βλέπετε αποκλειστικά και μόνο και με μεγάλη αυστηρότητα το θέμα της δημοσιονομικής πειθαρχίας και της πειθαρχίας όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά δεν εστιάζεστε καθόλου ε, στην κακή διαχείριση ε, και αντιθέτως ε, με την απόφασή σας υφίστανται κυρώσεις οι εργαζόμενοι. Η κατάσταση αυτή είναι απαράδεκτη. Καταλαβαίνουμε βεβαίως ότι η δημοσιονομική πειθαρχία και η πειθαρχία όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις είναι σωστή, αλλά θα πρέπει να δούμε τη γενικότερη εικόνα. Ευχαριστώ πολύ, Ελεονόρα. Ναι, θα προσθέσω μόνο το εξή ε, γιατί συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπε ο συνάδελφος Μάρκο Βάλλη. Ε, το μόνο που μπορώ να πω εδώ και να προσθέσω, να προσθέσω είναι ότι δεν είχαμε καμία διαφάνεια ε, και είχαμε μεγάλες δυσκολίες για να έχουμε πρόσβαση στα έγγραφα. Στο, ε, πρέπει να σας πω επίσης ότι ούτε εμείς ούτε οι εργαζόμενοι ε, στην εταιρεία είχαν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα έγγραφα ε, στον Δήμο του Μιλάνο Θεωρούμε λοιπόν ότι αυτό είναι ιδιαίτερο ανησυχητικό. Η, κατά την δική μου άποψη θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά αυτή έτσι ώστε να δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε σχετικά με την έρευνα αυτή, να κατανοήσουμε ποιος έχει την ευθύνη, κυρίως, ποιο, ε, κυρίως ποιος έχει την πολιτική ευθύνη για αυτήν την τόσο κακή διαχείριση. Ευχαριστώ. Η πρόεδρε, ευχαριστώ. Δεν βλέπω κανέναν άλλο. Ή μήπως παρέβλεψαν κάποιον. Καλά λοιπόν, επιστρέφω την, ε, το μικρόφωνο στον ε, ε, αναφερόμενο. Για δύο λεπτά παρακαλώ. Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Ε, ανησυχούν πολλοί οι εργαζόμενοι και θέλουν δύο πράγματα να απαντήσει άμεσα η Κομισιόν. Ε, πρώτον, εάν αυτό το, αυτή, η, το περιβόητο πρόστιμο ε, ισχύει ακόμα ή όχι ε, αν έχει ακυρωθεί ή όχι. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, ε, υπάρχει μία πρόθεση διαδικασίας επί παραβάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την εταιρεία Airport. Ε, ρωτώ λοιπόν, εάν έχει καταργηθεί το πρόστιμο με την δημιουργία της νέας εταιρείας και επίσης εάν υπάρχει νέα πρόθεση νέου προστίμου, υποβολής νέου προστίμου στην νέα εταιρεία. Πριν από δύο χρόνια έπρεπε να αποφανθεί το δικαστήριο του Λουξεμβούργου Λουξεμβούργου επ' αυτού ε, και ρωτώ την Επιτροπή γιατί δεν έχουμε πληροφορίες επ' αυτού. Το πρωτοδικείο του Λουξεμβούργου έχει ήδη πάρει απόφαση. Actually, that Δεν έχω κανένα άλλο εγγεγραμμένο ε, συνάδελφο. Νομίζω όπως πρότεινε ο κύριος Γιάρ, να κρατήσουμε την αναφορά ανοιχτή, να αναμείνουμε την τελική απάντηση και αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πάντως αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να γράψουμε επιστολή στον Δήμο Μιλάνου για να προτείνουμε να βρεθούν καλύτερες βιώσιμες λύσεις προς το συμφέρον των ε, ε, εργαζομένων αλλά και των επιβατών του αεροδρομίου. Νομίζω με τον τρόπο αυτό μπορούμε να δείξουμε ότι όντως ε, εγκύπτουμε στο θέμα τους ακόμη και αν βεβαίως πρόκειται για υπόθεση η οποία εκκρεμεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Αλλά με τον τρόπο αυτό να δείξουμε ότι και εμείς οι Ευρωβουλευτές ενδιαφερόμαστε πολύ για τα όσα συμβαίνουν εκεί. Συμφωνείτε? Ευχαριστώ πολύ. Ελεονόρα, εσείς να προσθέσουμε στην επιστολή, να τονίσουμε δηλαδή την ανάγκη διαφάνειας και πρόσβασης σε πληροφορίες και από τους εργαζόμενους και από τους πολίτες για το συγκεκριμένο θέμα. Και μήπως μπορεί να απαντήσει συντόμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ο αναφερόμενος έθεσε και μια-δυο απλές ερωτήσεις. Επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει συντομότατα στον αναφερόμενο. Βεβαίω, απαντάει η Επιτροπή. Ορίστε παρακαλώ. Πρώτον, εάν εκκρεμεί ακόμα η διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Επ' αυτού μια διασάφηση. Δεν πρόκειται για διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Πρόκειται μάλλον για απέτηση επιστροφής αδικαιολογήτως καταβληθέντων για να επανέλθουμε στην κατάσταση η οποία υπήρχε πριν από την καταβολή των επιδοτήσεων. Δηλαδή, για να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς με τον τρόπο ώστε να μπορούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους και οι ανταγωνιστές της συγκεκριμένης εταιρείας. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει βεβαίως και σε βιώσιμες θέσεις απασχόλησης. Άρα δεν πρόκειται για διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Τώρα, για την διαδικασία απαιτήσεω των αχρηστών καταβληθέντων. Ναι, αυτή εκκρεμεί. Συνεχίζεται δηλαδή. Εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση της Επιτροπής να απαιτήσει επιστροφή των καταβληθέντων ποσών. Γνωρίζει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Sea Handling βρίσκεται σε διαδικασία πτωχεύσεως. Και τώρα έχει αναλάβει η Airport Handling, η οποία εξακολουθεί να είναι ενεργός. Είπα και πριν ότι ξεκίνησε νέα διαδικασία η οποία εξετάζει εάν η airport handling απολαμβάνει πλέον το πλεονέκτημα που προσφέρουν εκείνες οι μη νόμιμα καταβληθήσεις επιδοτήσεις. Αυτή η διαδικασία κρεμεί και θα ληφθεί εν τέλει απόφαση επί της ουσίας, αν όντως υπάρχει τέτοιο πλεονέκτημα ανταγωνισμού ή όχι. σχετικά με το ερώτημα για την διαφάνεια. Η τυπική διαδικασία που διεξάγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποκαθιστά την διαφάνεια με την έννοια ότι και όσοι συμμετέχουν στην αγορά και ε, το κράτος της Ιταλίας και η περιφέρεια όλα θίγονται από αυτά. Οι γνωμοδοτήσεις τις οποίες έχουμε λάβει από την c Ending αλλά και από την Ιταλική Δημοκρατία και από άλλους φορείς θα εξεταστούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να λάβει την τελική απόφαση. Και μια τελευταία φράση για την εφαρμογή του δικαίου επιδοτήσεων ή ενισχύσεων καλύτερα. Κατανοώ ότι μπορεί να ανησυχούν πολύ ορισμένοι για τις αρνητικές επιπτώσεις από την πτώχευση της ε, Sea Handling, ωστόσο το δίκαιο των ενισχύσεων δεν μπορεί να εγκύψει στην προκειμένη περίπτωση, στην προκειμένη υπόθεση μάλλον. Ο σκοπός του δικαίου αυτού είναι να αποκαταστήσει τον ε, ανταγωνισμό. Σας ευχαριστώ πολύ για την ε, πρόσθετη αυτή εξήγηση. Άρα, επαναλαμβάνω, διατηρούμε την αναφορά ανοιχτή, αναμένοντας πλήρη επίσημη απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αποστέλουμε επιστολή στον Δήμο Μιλάνου, τονίζοντας ιδιαίτερα την κατάσταση των εργαζόμενων. Έτσι θα προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήλθατε εδώ. Και θα εξακολουθούμε να, να παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Η επόμενη τώρα διαφάνεια αναφέρεται στην ε, ποιότητα του πόσιμου νερού στην, ε, στην χώρα των Βάσκων. Ε, νομίζω ότι ο αναφερόμενος είναι παρόν. Θα σας δώσω τον λόγο για πέντε λεπτά. Μάλιστα νομίζω ότι υπάρχει και σχετικό βίντεο. Where is, where is the petitioner? Πού κάθεται παρακαλώ αναφερόμενος. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Έχετε τον λόγο κύριε για πέντε λεπτά.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 Hainbat analisi egin ostean, kutsaduraren jatorria oiolako urtegia dela ondorioztatu zuten. Orduz geroztik, oiolatik datorren ur hornidura hainbat aldiz eten dute, baina herritarrek lindanos kutsatutako ura erabiltzen jarraitu dute tarte luzeetan. Aquí abajo tenemos la escorrentía de la Gorriga, ¿eh? que recoge el agua del arroyo Ángela, que es por donde entra el HCH en el pantano de Oyola, que lo tenemos aquí enfrente, en la Diputación. Εδώ βλέπετε στην περιοχή μας την ε, λεκάνη υδατός η οποία έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια δεν ε, είναι μολυσμένη από λινδάνιο. Άλλοι μας λένε όπως οι αρχές ότι δεν έχει μολυνθεί και είναι πόσιμο το είδες. Αυτό το οποίο όμως είναι σαφές είναι ότι όσο και αν είναι σε μηδενικά επίπεδα η μόλυνση από το λινδάνιο, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Έχουμε εδώ να κάνουμε εξαιτία αυτής της μόλυνσης στην περιοχή αυτή με μεγάλες ποσότητες οι οποίες δεν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 ευχαριστήσω που μας επιτρέψετε να έρθουμε εδώ και να ακούσετε τις ε, αξιώσεις που έχουμε και να ακουστεί η φωνή μας. Είναι η τρίτη φορά που ερχόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θα μακρηγορήσω, διότι συνοπτικά έκανε την παρουσίαση το βίντεο. Με σαφήνεια και βεβαίως σε όλα τα έγγραφα που έχετε, έχετε που σας έχουν αποστολή, έχετε τις εκθέσεις και τις απαιτήσει μας. Αυτό που θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Επιτροπή σας είναι να προσέξετε ιδιαίτερα το θέμα αυτό, ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιμείνει σε όλα τα θεσμικά μας όργανα, σε κεντρικό επίπεδο και σε επίπεδο αυτονομιών για να συνεργαστούν οι πάντες ώστε να ευρεθεί λύση. Δεν θα πρέπει να πετάει το μπαλάκι ο ένας τον άλλο στην Ισπανία λέγοντας ότι αυτός που πρέπει να επιλύσει το πρόβλημα και να ενεργήσει είναι ο άλλος. Διότι έτσι δεν φτάνουμε πουθενά. Κάνουμε λοιπόν έκκληση σε εσά και ζητούμε με οκτώ σημεία σαφή το εξή. Πρώτα απ' όλα να εντοπιστούν όλες οι, αιτίες, οι Με σφαιρικό τρόπο να επιληθεί το πρόβλημα. Να μην και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει κανείς να έχει πόσιμο είδος να ευρεθούν ποιες είναι οι περιοχές, ποτάμια, οι λίμνες, τις οποίες υπάρχουν αυτές οι οσίες που μολύνουν το είδωρο. Να υπάρξει καθαρισμός αυτών των περιοχών, να γίνουν έρευνες, να αποδοθούν ευθύνες που να ανταποκ... πολιτικές και διοικητικές και να δοθούν τα απαραίτητα κονδύλια ώστε όλες αυτές οι δράσεις που προανέφερα να γίνουν πραγματικότητα και τελικά να εγγυηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θα υπάρχει πλήρης διαφάνεια σε ό,τι γίνει και ότι θα συμμετάσχουν όλοι οι πολίτες διότι όλο μαζί, μόνον όλοι μαζί, όλες τα όργανα σε εθνικό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να εργαστούμε από κοινού για να εξεύρουμε λύση στο πρόβλημα. Σας ευχαριστώ. Έχουμε πάρα πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη και είμαστε φορτωμένοι πολύ. Πρέπει να σας διακόψω και να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να περάσω προς την Επιτροπή. Ο κύριος Γκόμες είναι μαζί μας, εκ μέρους της Επιτροπής. Του δίνω αμέσως το λόγο για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως μπορούσατε να δείτε στο βίντεο, αυτή η αναφορά αφορά την μόλυνση από το λινδάνιο, που είναι η εμπορική ονομασία του ζυζανιοκτόμου που είναι τόσο πολύ επικίνδυνο για την ουσία, στα είδα τα, οποία ε, μαζεύονται για να προμηθευτούν διάφοροι δήμοι και μικρές πόλεις στην περιοχή της Όλα τα θέματα που αφορούν τον κίνδυνο για τη δημόσια υγεία είναι θέμα προτεραιότητας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίω για, την για τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντο. Όταν ενημερωθήκαμε για το θέμα αυτό είπαμε ότι θα κάνουμε έρευνα ώστε να μπορέσουμε σε επαφή με τις ελληνικές αρχές να δούμε αν εφαρμόζεται σωστά το ευρωπαϊκό δίκαιο στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα πρέπει να διευκρινίσω παρόλο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί μόνο να παρέμβει σε θέματα τα οποία καλύπτονται από το κοινοτικό δίκαιο αλλά δεν έχει αρμοδιότητες για να παρέμβει σε οποιοδήποτε άλλο θέμα το οποίο δεν το θεσπίζει η κοινοτική νομοθεσία. Κατά συνέπεια, έγινε η έρευνα αυτή όσον αφορά την εφαρμογή προδιαγραφών και κανόνων που συμπεριλαμβάνονται στο κοινοτικό δίκαιο σε σχέση με την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είδε ότι όντως εφαρμόστηκε σωστά η 9883 οδηγία για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Αυτή η οδηγία δίδει τις παραμέτρους ώστε το νερό το οποίο ε, προβλέπεται για ανθρώπινη χρήση είναι καθαρό νερό και πόσιμο. Τώρα να αποφασίσουμε εάν αυτά τα ύδατα ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτών των παραμέτρων έγιναν μετρήσεις στην βρύση, στο νερό που βγαίνει από την βρύση, το οποίο καταναλώνουν οι αρχές στην Ισπανία όντως αναγνώρισαν ότι είχε συμβεί ένα επεισόδιο μόλυνσης του 2008, τον Ιούλιο του 2008, συγκεκριμένα από Λινδάνιο και εκείνη την ε, εποχή έλαβαν τα, κατά την άποψή τους, κατάλληλα μέτρα για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα μόλυνσης του είδου. Σύμφωνα με τις προφορίες που μας διαβίβασαν, αυτή η περίοδος μόλυνσης σε ανώτατο όριο ήταν τριμηνιαία περίοδος. Μεταξύ λοιπόν των δύο μετρήσεων και δειγμάτων που ελήφθησαν, ορίστηκε αυτή η χρονική περίοδος, απαγορεύθηκε η χρήση αυτού του νερού ως πόσιμο και χρησιμοποιήθηκαν άλλες φυσικές πηγές. Οι αρμόδιες αρχές Επίσης είδαν ποιες ήταν οι αιστείες μόλυνσης. Αυτό ήταν κάτι που γινόταν και από προηγούμενα χρόνια, αλλά έγινε πιο εντατική έρευνα, ώστε να μπορέσουν να ε, τερματίσουν οποιαδήποτε τέτοια αιστεία μόλυνσης από Λινδάνιο. Εκ των υστέρων, τα αποτελέσματα των αναλύσεων που έγιναν για να μπορέσει να ξαναχρησιμοποιηθεί το νερό σε αυτή την λιμνοδεξαμενή στην Ογιόλα. Όλες οι μετρήσεις, επαναλαμβάνω, ήταν σύμφωνες με τις μετρήσεις που προβλέπει η σχετική οδηγία, η οποία θεσπίζει όσο όριο 0,1 μικρογραμμάριο ένα λίτρο για τα ζυζανιοκτώνα σαν το και 0,5 για το σύνολο των άλλων εντομοκτώνων και ζυζανιοκτώνων. Σύμφωνα με τα παρόντα αποτελέσματα δεν ε, ξεπερνιέται για το λινδάνιο το 0,01 μικρογραμμάρι για το λινδάνιο καθώς ε, και ε, τα ανώτατα όρια γενικότερα για όλες τις επιβλαβείς ουσίες. Δηλαδή τα όρια είναι πολύ πιο κάτω από τα θεμητά. Οι αρχές στην Ισπανία μας είπαν ότι έκαναν επίσης ανάλυση κινδύνου για να δουν κατά πόσον αυτό το συγκεκριμένο ε, πρόβλημα αποτελούσε κίνδυνο για την δημόσια υγεία και το συμπέρασμα ήταν ότι κατά το όριο η έκδοση σε αυτό το υψηλότερο ποσοστό ήταν τρεις μήνες, αλλά δεν ήταν το ποσοστό τόσο πολύ υψηλό ώστε να υπάρξει για τρεις μήνες κίνδυνος. Και βεβαίως έγινε η σχετική ενημέρωση σε όλους τους κατοίκους όταν ε, ε έμαθαν και ποιες ήταν ενδεχομένως οι πηγές μόλυνσης. Άρα πιστεύουμε ότι δεν έγινε παραβίαση των υποχρεώσεων της σχετικής οδηγίας για την ποιότητα του πόσιμου ύδατος. Η Επιτροπή όχι μόνο λοιπόν έκανε έρευνα στην, για την ποιότητα του νερού που μετρήθηκε ε, ώστε να ξέρουμε τι ακριβώς έπιναν οι πολίτες, αλλά είδαμε και στην οδηγία πλαίσιο του 2260 το ότι θα πρέπει σε πριν από το 2011 να υπάρχουν, γίνονται σεβαστές κάποιες σχετικές ε, παράμετροι για το πόσιμο είδος. Η καλή ποιότητα της χημικής ανάλυσης καθορίζεται από τις ε, σχετικές παραμέτρους και στη συγκεκριμένη περίπτωση εφαρμόστηκε για το Λινδάνιο. Η Επιτροπή επίσης ανέλησε την απάντηση των αρχών των Ισπανικών και επαλήθευσε ότι οι αρχές αυτές όντως αναλύουν τα, σε τακτά διαστήματα τα νερά στην περιοχή αυτή και υπάρχει πλήρης συμμόρφωση με την σχετική οδηγία. Εξάλλου, το ε, σχέδιο ε, της περιοχής λεκάνης απορροής του ποταμού της περιοχής καθόρισε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση στην Ογιόλα προβλέπεται ένα σχέδιο δράσης ώστε να επιληθεί το πρόβλημα που δημιουργείται στην περιοχή Θαϊθάμπαλη με το λινδάνιο και προβλέπεται και κονδύλι σχετικό 50.000 ευρώ. Η Επιτροπή λοιπόν δεν μπόρεσε να διαπιστώσει ότι υπάρχει παράβαση της σχετικής οδηγίας και θεώρησε ότι δεν θα πρέπει να συνεχίσει την έρευνα δεδομένου ότι έτσι όπως προβλέπει το κοινοτικό δίκαιο ε, πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εκ μέρους των ε, Ισπανικών υπεύθυνων αρχών. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχουν οι συνάδελφοι τώρα. Ο κύριος Χουάρεγη πρώτα απ' όλα. Συγγνώμη που δεν προσφέρω σωστά το όνομά σας, έχετε το λόγο. Καλά, καλά το είπατε, καλά το είπατε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αυτό το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι... Ωραία, το ότι ο κίνδυνος τη δημόσια υγεία είναι κάτι που ανατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θεωρεί ότι έγιναν ε, σεβαστές οι διάφορες παράμετροι. Δεν εξηγούνται όμως κάποια πράγματα και για τους πολίτες ο τρόπος τον οποίο ενήργησαν οι αρχές δεν ήταν ο καλύτερος και ο πιο κατάλογος. Οι πολίτες πιστεύουν ότι παραμένει το πρόβλημα και όχι μόνο η αιστεία της μόλυνσης παραμένει, κατά την άποψή μου θα πρέπει να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις αρμόδιες αρχές να συνεργαστούν μεταξύ τους, κάτι το οποίο δεν το κάνουν, δεν το κάνουν καθόλου, χάνουν χρόνο και δημιουργούν κάποια ε, αισθήματα ε, αβεβαιότητας και έννοιας για τους πολίτες, θα πρέπει με τρόπο συντονισμένο να εργαστούν οι πάντες, ακόμη και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών κινημάτων και όλοι οι υπεύθυνοι φορείς, ώστε να μπορέσει να επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Δεν σημαίνει αυτό μόνο στην περιοχή του Ογιόλα, αλλά θα δείτε αργότερα και στο ποτάμι Γαλιέγο και σε άλλες περιοχές της Ισπανίας τουλάχιστον. Θα πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να επιληφθεί του όλου θέματος. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ζητηθεί να γίνει μια νέα ευρωπαϊκή έκθεση επί αυτού του θέματος για να είμαστε σίγουροι ότι ενεργούμε σωστά. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σεμπαστία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται τη στιγμή κατά την οποία το νερό που κατανάλωναν οι πολίτες της περιοχής που προμηθεύονταν από το Ογιόλα δεν ανταποκρίνονταν στα κανόνες υγιεινής όταν, σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Έχουμε όμως εδώ προηγούμενο, είναι προηγούμενο του τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Και όπως ελέγχθη, δεν μπορούμε να επαληθεύσουμε το ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη που είναι η αιστεία της μόλις. Το πρόβλημα του λινδανίου είναι πάρα πολύ σοβαρό σε πολλές περιοχές της Ευρώπης. Στην περιοχή του Ογιόλα και της λεκάνης αυτής έχει προσθέμενη αξία γιατί ξέρουμε περίπου που ε, περνάει αυτό το, το λινδάνιο που αφέθηκε και που φιλτράρεται. Τα ξέρουμε όλα αυτά. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να κάνει στου αρμόδιους φορείς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να μπορεί να εξασφαλίσουν ότι δεν θα υπάρξει τέτοιου είδου περίπτωση στο μέλλον. Και ξέρω ότι δεν μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό γιατί δεν ξέρουν που βρίσκεται η αστεία τη μόλυνσης. Θα πρέπει λοιπόν να συμμετάσχει στην επίλυση του θέματος αυτός η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συντονισμό όπω ζητούν οι κάτοικοι τη περιοχή. Και το θέμα νομίζω ότι δεν λύνεται με συγκεκριμένου ελέγχους κάποιες μέρες. Η λύση είναι πλήρης όταν ξέρει κανείς που είναι η αστεία της μόλυνσης και όταν σταματήσει να υφίσταται τέτοιου είδους ε, αιστεία. Κατά συνέπεια, πιστεύω ότι έχουμε ακόμη πολλή δουλειά μπροστά μας και αυτό το προηγούμενο μας καταδεικνύει ότι συνεχίσει να υπάρχει κίνδυνος. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη, δεν σας βλέπω καλά, γιατί πέφτει ο ήλιος ε, στα μάτια μου. Ε, κύριε Ελβιόλα, δεν ε, είδα που ζητήσατε το λόγο. Σας, σας τον δίνω πάντως. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι εδώ έχουμε μία σαφή περίπτωση μόλυνσης ε, του περιβάλλοντος και απειλής κατά της δημόσιας υγείας. Εδώ μιλάμε για τοξικά κατάλοιπα, ε, για, μιλάμε για μολυσμένα νερά, μιλάμε για, ε, για ζώα τα οποία μολύνονται με επιμόλυνση και των ανθρώπων. Θεωρούμε ότι οι δημόσιες αρχές δεν αντιμετώπισαν σωστά τα πράγματα, ούτε από την πλευρά της κεντρικής κυβέρνησης, ούτε και από την πλευρά της αυτόνομης κυβέρνησης. Γι' αυτό λοιπόν ε, μάθαμε αυτά που μας είπαν ε, οι αναφερόμενοι και κατά αυτή την έννοια πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, να υπάρξει έκθεση από, πλευράς, από ευρωπαϊκής πλευράς για το θέμα αυτό, για τον Παρακάλντο, για, την, για τον ταμιευτήρα του ΟΙΟΛΑ και έτσι ώστε να προβλέψουμε και να αποφύγουμε παρόμοιες καταστάσεις στην, Ευρώ... στην υπόλοιπη Ευρώπη. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα του Λινδανίου και ε, πιστεύω ότι τέτοιου είδους αναφορές θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, διαβιβάζονται και στην ΕΜΒΗ, στην Επιτροπή Προστασίας του ε, Περιβάλλοντος, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσον υπάρχει παραβίαση όσον αφορά την ποιότητα, την οδηγία ποιότητα των νερών κτλ. Να οι ανοιχτή λοιπόν αυτή η αναφορά. Thank you very much. Now I can really assure you that I see everyone perfectly. Τώρα είμαι πάρα πολύ καλά, σας βλέπω όλους ε, τέλεια, αλλά βεβαίως αφήσαμε και τον ήλιο έξω από την αίθουσα. Δεν βλέπω να ζητά κάποιος άλλος το λόγο. Α, ο κύριος Καλβέτ και ο κύριος Λαφριέ. Κύριε Καλβέτ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό το πρόβλημα με το λινδάνιο που το ζούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αλλά κυρίως στην περιοχή της Αραγωνίας, εκεί γεννήθηκα στην Ισπανία, μπορεί να είναι μια πάρα πολύ σαφής περίπτωση ευτυχούς παρέμβασης της Επιτροπής μας από την στιγμή που εμείς δεν είμαστε γραφείο παραπώνων, αλλά νομοθέτες, πολιτικοί και μπορούμε να πάρουμε κάποιες πρωτοβουλίες. Ελπίζω ότι ποτέ δεν υπήρξαν θύματα από το λινδάνιο, αλλά όντω πρόκειται για κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ω ουσία επικίνδυνη. Πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα. Το ότι πήρανε μία πρωτοβουλία οι Ισπανοί δεν μειώνει το πρόβλημα. Πιστεύω ότι η Επιτροπή μας και επαναλαμβάνω αυτό που είπα, να ζητήσουμε και από την ΕΜΒΗ και από όλους τους υπεύθυνους να κάνει μία μελέτη για τους κινδύνους που απορρέουν από την πρόσληψη κάποιου τέτοιου είδους ε, δηλητηρίου όπως είναι το λινδάνιο και βεβαίως να δοθούν και τα κατάλληλα κονδύλια. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να ζητήσουμε, επαναλαμβάνω, και κονδύλια. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίως πρέπει να πω ότι ευτυχώς χτύπησε το καμπανάκι κινδύνου στην Ισπανία. Πιστεύω όμως ότι η επικινδυνότητα είναι πάρα πολύ σημαντική από το Λινδάνιο και δεν θα πρέπει να την ε, παραγνωρίσουμε. Eh, eh, Πιστεύω λοιπόν ότι μία πρωτοβουλία κοινοβουλευτική προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν κάτι το πολύ θετικό και βεβαίως να διατεθούν επαναλαμβάνω και τα κατάλληλα κονδύλια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Λαμπριέ. Merci, Madame la σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και τι ωραία που προφέρατε το όνομά μου, εξαιρετικά γαλλικά. Να υπενθυμίσω ότι εδώ βρισκόμαστε στην Επιτροπή Αναφορών ε, όπου ε, ασχολούμαστε με ένα συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο αφορά την Ισπανία. Άκουσα τις εξηγήσεις και του αναφερομένου και της Κομισιόν. Σύμφωνα με τα ε, στοιχεία τα οποία μας έχουν, μας έχουν υποβληθεί δεν υπάρχει παραβίαση κανενός ευρωπαϊκού ενωσιακού κειμένου ε, και ε, λήφθησαν τα μέτρα έτσι ώστε να σταματήσει μία ρήπανση η οποία αν κατάλαβα καλά έλαβε χώρα το 2008. Ε, υπενθυμίζω λοιπόν ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση όλοι έκαναν τη δουλειά που έπρεπε να κάνουν. <clears throat> Ζητώ λοιπόν, ζητώ λοιπόν σαν μέλος της Επιτροπής Αναφορών να διαπιστώσουμε ότι όλοι έκαναν καλά τη δουλειά τους, να ε, λάβουμε υπόψη μας ε, ότι ε, τα στοιχεία ελήφθησαν σωστά υπόψη, να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι ότου μελετηθούν και τα νέα στοιχεία και μετά, κυρία Πρόεδρε, Νομίζω ότι μπορώ να καλέσω τους ε, συναδέλφους που δεν έρχονται κάθε φορά ε, στην Επιτροπή Αναφορών να ασχοληθούν στην Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος με ένα ευρύτερο ζήτημα που είναι αυτό της ρήπανσης από λινδάνιο ε, γιατί εδώ εμείς δεν είμαστε επιτροπή που ασχολείται με περιβαλλοντικά θέματα, ούτε μπορούμε να παίξουμε το ρόλο αυτής της ε, επιτροπής και να την υποκαταστήσουμε. Είμαστε επιτροπή αναφορών και δεν είμαστε αρμόδιοι ε, καθήλυν και επομένως μπορούμε να διαβιβάσουμε σε αυτούς το θέμα. Εμείς είμαστε η Επιτροπή στην οποία απευθύνονται οι πολίτες όταν δεν έχουν άλλα μέτρα προσφυγής. Ε, εδώ διαπιστώνουμε λοιπόν ότι ο καθένας από τους εμπλεκομένους έκανε τη δουλειά που έπρεπε να κάνει και τελεία. και βεβαίως ε, ως αναπληρωτής, ε, ε, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Αναφορών δεν έχω κανένα πρόβλημα να είμαι παρόν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος όταν θα μελετήσουν το θέμα αυτό. Επαναλαμβάνω λοιπόν την πρότασή μου μέχρι ότου έχουμε τα αποτελέσματα των συμπληρωματικών αναλύσεων για τη συγκεκριμένη περίπτωση να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά. Όσον αφορά τα γενικότερα ζητήματα για Λινδάνη δάνειο κλπ. Ε, ε, πλήρως εμπιστεύομαι τους συναδέλφους της Επιτροπής Περιβάλλοντος και δεν θέλω να ασχοληθώ με θέματα που είναι δικιά τους αρμοδιότητας. Η κυρία Αγιάλα Σέντερ παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί τη ότι δέχεστε να μιλήσουμε και εμείς ε, οι βουλευτές που δεν είμαστε μέλη της Επιτροπής σας. Και διότι προσπαθούμε όλοι μαζί να κάνουμε κάτι σαν ένα πρώτο βήμα για να επιληθεί το πρόβλημα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το πρόβλημα αυτό που σας ε, υπέβαλε ο αναφέρον. Πολλές φορές έχει περάσει ε, και από την ε, Επιτροπή Ελέγχου του Υπουργού την δική μας έχουν περάσει τέτοιου είδους θέματα όπως αυτά και έχουν ζητηθεί και κονδύλια. Υπάρχουν δύο-τρία παραδείγματα ήδη τέτοιες ε, είδη τρόπου ε, ανταπόκριση εκ μέρου μας και νομίζω ότι εκτός από αυτά τα οποία είπε η Επιτροπή θα πρέπει να ανοίξει και ένα φάκελο που έχει να κάνει και με την ε, μόλυνση του εδάφου στις περιοχές αυτές διότι πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και χρόνια θα έπρεπε να το έχει κάνει και προς το παρόν αφήνει τα πράγματα ως έχουν. Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο όμω δεν αφορά μόνο την Ισπανία, όπω συγκεκριμένη περίπτωση με το Λινδάνιο, σε άλλε χώρε. Δεν ξέρω στη Γαλλία τι γίνεται, στη Γερμανία επίση, κοντά στο Αμβούργο. Αρκετού θέματα και παρά το γεγονό ότι ακόμη δεν έχουν δοθεί οι πλήρεις λύσεις και δεν μπορούν να δοθούν λύσεις για τα θέματα αυτής της μόλυνσης, θα πρέπει να γίνει μια σωστή μελέτη για να δούμε περί τίνος ακριβώς πρόκειται για να χαρτογραφήσουμε και κατά κάποιο τρόπο την ε, κατάσταση που δημιουργείται από την χρήση του λινδανίου και άφησε και την, το αποτύπωμά του, το αρνητικό, και σε άλλες περιοχές της Ευρώπης. Για να μπορέσουμε με ένα σχέδιο δράση από κοινού να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημα της χρησιμοποίησης ε, μία ουσίας επικίνδυνης που μολύνει πολύ και δεν βιοαποδομείται εύκολα. Μένει για πάρα πολύ καιρό στις περιοχές που έχει μολύνει και δεν υπάρχει ούτε μεγάλη, ε, δεν έχουν δοθεί ούτε πολλά κονδύλια, ούτε έχουν γίνει μελέτες για να δούμε πώς μπορούμε να απαλλαγούμε αυτό το θέμα. Και η Γαλλία Ξέρουμε ότι έχει το ότι έχει πολιτική υπομόλυνση, ξέρουμε ότι υπάρχει τεχνογνωσία και από άλλε χώρε για να μπορέσει να καθαριστεί μια περιοχή. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε κάτι και η Επιτροπή θα πρέπει να ζητήσει να γίνει αυτή η χαρτογράφηση, όπως σας είπα, των μολυσμένων περιοχών από αυτή την χημική ουσία και να δούμε πώς ε, οι γεωργικές ε, η γη η οποία ε, έχει γεωργική χρήση καθώς και το νερό το πόσιμο μπορούν να απαλλαγούν από αυτή την τόσο μολυσματική ουσία. Ξέρουμε πόσο έχει συνεισφέρει και το ρίτσε στο να εντοπιστούν τέτοιου είδους ουσίες. Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκε ο κατάλογος των ομιλητών. Κύριε Βελάσκο, μπορείτε να κλείσετε εσείς ε, συνοπτικά σε λιγότερο από δύο λεπτά. Να προσθέσετε κάτι. Θα ήθελα να διευκρινίσω το εξής. η ενημέρωση και τα έγγραφα τα οποία έστειλε η τοπική μας αυτοδιοίκηση ή η κεντρική μας κυβέρνηση είναι λίγη, ζητήσαμε αυτά τα σχετικά έγγραφα να μας διαβιβαστούν και σε μας. Ακόμη δεν τα έχουμε λάβει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε παρουσιάσει στην Επιτροπή. Πράγμα το οποίο είναι ενδιαφέρον στην έκθεση είναι να δούμε ε, τι έγινε για να μπορέσουμε να απαλλαγούμε από την μόλυνση όταν είπε ότι κλείσαν δύο χωματερές. Αυτό έγινε το 2012, αλλά έχουμε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο το 2014 που έχουμε 250 νανογραμμάρια ε, λιντανίου αναλύτρου. Αυτό καθιστά απόλυτα σαφές ότι δεν επιλύθηκε το πρόβλημα, ότι ακόμη δεν γνωρίζουμε από πού προέρχεται αυτή η μόλυνση, εάν ξέρουμε από πού προέρχεται, δεν λαμβάνονται τα κατάλληλα προστατευτικά μέτρα, ώστε το ζωικό κεφάλαιο, το οποίο είναι στην περιοχή, ούτε να πίνει νερό, ούτε ζωοτροφές οι οποίες έχουν μολυνθεί. Πιστεύω λοιπόν ότι εάν δεν μπορεί κάποιος στο επίπεδο ε, εθνικό να λυθεί το πρόβλημα, μόνο με τη συνδρομή όλων και με συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων φορέων με την κυβέρνηση θα μπορέσει να λυθεί. Γι' αυτό ζητούμε συντονισμό και συνεργασία. Πρέπει να σας πω ότι ε, προσκλήθηκε και αντιπροσωπεία της ε, χώρας των Πάσκων. Ε, δεν είναι κάτι καινούριο σε αυτή τη συνεδρίαση, δεν είναι καινούριο αυτό και ήδη το 2014 τον Μάρτιο η Επιτροπή μας ε, έστειλε επιστολή ε, στις ε, τοπικές αρχές των υδάτων καθώς επίσης και στα δημοτικά συμβούλια έτσι ώστε να, έχουν, ε, να ε, έχουμε πληροφορίες σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, μονάχα απήντησε η αρχή της κεντρικής κυβέρνησης λέγοντας ότι θα μας απαντήσει αργότερα εντελεχώς αλλά δεν λάβαμε ποτέ αυτή την εντελεχή απάντηση. Κοιτάξτε, ε, νομίζω ότι προς το καλό όλων, καλό είναι να γνωρίζουμε ποια είναι η αιστεία της ε, μόλυνσης, γιατί φαίνεται ότι αυτό το αγνοούν όλοι. Νομίζω ότι αγαπητοί συνάδελφοι έχετε απόλυτα δίκιο, θα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά και να επιμείνουμε ε, στέλνοντας ε, εκ νέου επιστολή στην ε, αρμόδια αρχή της χώρας των Βάσκων έτσι ώστε να, έχουμε, να λάβουμε τις απαραίτητες πληροφορίες, να καταλάβουμε πού είναι η πηγή γιατί εδώ μιλάμε για ένα παραστοκτόνο το οποίο είναι εξαιρετικά επιβλαβές για την ανθρώπινη υγεία. Επομένως, το αφήνουμε ανοιχτό και το θέμα αυτό αλλά και το επόμενο. Ε, τα στέλνουμε, τα προωθούμε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος γιατί είναι δικιά τους αρμοδιότητα να δουν πώς θα προχωρήσουν. Εμείς όμως, εμείς όμως θα τους στείλουμε ε, μία επιστολή μέσω της οποίας θα συστήνουμε ε, να μελετήσουν ευρεθώς το θέμα. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη αφορά το ίδιο πράγμα, αλλά από τη στιγμή που παρίστανται ε, και αναφερόμενοι από την Ιρλανδία και έχουν ε, χρονικό όριο πολύ σφιχτό γιατί έχουν ε, μία πτήση για να επιστρέψουν στην Ιρλανδία σε λίγο. Θα αντιστρέψουμε λίγο την σειρά και επομένως θα δώσουμε αμέσως το λόγο ε, στους αναφερόμενους του σημείου 11 μπορείτε να συμφωνήσετε συνάδελφοι. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Αυτό που θα κάνουμε λοιπόν τώρα είναι ότι θα ασχοληθούμε με την 1674 ε, του 2013 του Πίτερ Μακιού και μετά την 1022 του 12 επίσης Ιρλανδική ειδική ε, περίπτωση σχετικά με εσφαλμένη εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεων για τα συστήματα ενιαίας ενίσχυσης αναγεωργική γνωμοδότηση. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Πίτερ Μακχιού για πέντε λεπτά maximum. In Καλώς ήρθατε, σας είδα, είσαστε εδώ στο μέσον και παρακαλώ πολύ, ε, περιμένουμε να σας ακούσουμε. Hello. Uh, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε που μας δίνετε την δυνατότητα ε, να μιλήσουμε τώρα και όχι σύμφωνα με την αρχική ημερήσια διάταξη. Ε, εμείς ε, εκπροσωπούμε εδώ τον αναφερόμενο ε, Πίτερ Μακιού γιατί είναι 82 χρόνων και σε αναπηρικό καρότσι και δεν είχε τη δυνατότητα να είναι εδώ. Σας διαβάζω λοιπόν τι θα έλεγε. Σας ευχαριστώ πολύ αγαπητά μέλη της Επιτροπής Αναφορών για την δυνατότητα που μου δίνετε να, να, σας, να απευθύνω το λόγο ενώπιόν σας. Λυπούμε πάρα πολύ που δεν είμαι σε θέση να ε, είμαι ε, παρόν. Ε, πρέπει να σας πω ότι δυστυχώς πριν από μερικά χρόνια είχα υποστεί ένα αγροτικό ατύχημα το οποίο μου άφησε πολλά προβλήματα, κυρίως δε έχασα το αριστερό μου χέρι. Πέρασα πολύ καιρό στο νοσοκομείο, στη διάρκεια του οποίου η ε, η σύζυγός μου ήταν αυτή η οποία είχε αναλάβει το θέμα. Ωστόσο από το 1993 ε, δεν ε, αισθανόταν καλά η σύζυγός μου και τελικά αναγκαστήκε να υποβληθεί σε εγχείρηση μερικής αφαιρέσεως στομάχου λόγω καρκίνου του στομάχου. Δυστυχώς επομένως από αυτή τη στιγμή και πέρα δεν είχε τη δυνατότητα να ασχοληθεί περισσότερο με την αγροτική μας εκμετάλλευση ε, και ε, απλώς προσπαθήσαμε να ε, την διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο μέχρι ότου να μεγαλώσει ο γιος μας. Το 1995 δυστυχώς αναγκαστήκαμε με βοηθούς και με εργαζόμενους να κρατήσουμε την αγρικία μας μέχρι να αρχίσει η σύζυγός μου να ξαναδουλεύει. Το 1997 ενταχθήκαμε στο ε, στο ε, πρόγραμμα ε, αγροτικής βοήθειας και εντωμεταξύ ο γιος μας πήγαινε στη σχολή γεωπονικής. Ωστόσο δεν καταφέραμε να κρατήσουμε τα ζώα μας παρά και τις αγελάδες μας, παρά κρατήσαμε μονάχα τέσσερα ζώα. Το 99 λοιπόν ε, πουλήσαμε ε, την εκτινοτροφική μας ε, μονάδα και η γυναίκα μου αντιμετώπισε ακόμα περισσότερα προβλήματα υγείας και έμεινε κατά 50% ανάπηρη. Ε, και ζητήσαμε επομένως ε, την ε, ενιαία πληρωμή αλλά την ενιαία γεωργική πληρωμή αλλά το θέμα είναι ότι στην ουσία φαινόταν να είναι πάρα πολύ μικρή η, η γεωργική μας εκμετάλλευση. Καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους αυτού του είδους η πληρωμή δεν είναι καθόλου δίκαιοι Ε, Στο το single farm payment ε, ε, κατέβηκε στα 186 ευρώ ανά ε, εκτάριο από το 2000 ε, μέχρι το 2002 όμως ε, εμείς ξαναδουλέψαμε την γεωργική μας εκμετάλλευση 100% και χωρίς να στηριζόμαστε καθόλου οικονομικά. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν ζητούμε καμία ελεημοσύνη, ζητάμε μονάχα να μας, να μας δοθούν αυτά τα οποία δικαιούμαστε μετά από πολλά χρόνια σκληρής δουλειάς ε, τώρα βρισκόμαστε στο 2016 τα, και τα έτη αναφοράς είναι τα έτη 2000-2002. Εμείς είμαστε μικροί γεωργοί ε, και επομένως ε, πιστεύω ότι θα πρέπει να βοηθηθούμε έτσι ώστε να μην τα χάσουμε όλα. Για μία ακόμα φορά πρέπει να σας πω ότι όσον αφορά την ενιαία πληρωμή και όσον αφορά τα όσα μας έχει απαντήσει μέχρι τώρα το Υπουργείο Γεωργίας βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και επομένως επομένως περιμένουμε να παραμείνει και σας ζητούμε να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά μέχρι ότου διαλευκανθεί η κατάσταση. Fine. Σας ευχαριστώ πολύ. Ας σχολιάσουν οι συνάδελφοι, διότι δεν υπάρχει εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσει, αλλά για άλλη Ιρλανδική αναφορά. Πέτερ Γιάρ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Τα όσα ανέπτυξε ο αναφερόμενος πράγματι οριοθετούν ένα πολύ δυσχερές πρόβλημα. Από την σκοπιά του νομοθέτη κάθε αλλαγή θα πρέπει να, υπάρχει, να, βασίζεται σε μια βάση. Και από τη δική μου εκλογική περιφέρεια τα γνωρίζω αυτά. Έχουν δοθεί δυνατότητες σε εθνικές αρχές να λαμβάνουν υπόψη τους ιδιαίτερα δυσχερείς περιπτώσεις. Ο λόγος για τον οποίο δεν έγινε στην προκείμενη περίπτωση ξεφεύγει από τα όσα γνωρίζω. Τα ίδια λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξετάσαμε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, λένε δώσαμε περιθώριο στις εθνικές αρχές. Από τα, από τα όσα άκουσα από το αναφερόμενο δεν κατανοώ γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν τα περιθώρια αυτά οι εθνικές αρχές θεωρώ ότι πρέπει να ξαναγράψουμε στις εθνικές αρχές της χώρας του και για να το πω πολύ στεγνά, οι εθνικές περιφερειακές αρχές έχουν ακριβώς αυτό το σκοπό να βοηθήσουν τους αναφερόμενους σε μια δύσκολη περίπτωση ασθενή ε, ο αναφερόμενο στην υπόθεση αυτή υπάρχει όμως και το φάρμακο. Γιατί δεν του χορηγήθηκε το φάρμακο δεν κατανοώ. Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η απάντηση. Πιθανώ να μπορεί να δώσει την απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι λέει ότι εμείς από την Ευρωπαϊκή Σκοπιά προβήκαμε στη μεταρρύθμιση και ψηφίσαμε του σχετικού νόμου. Η εφαρμογή στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να είναι έργο των εθνικών αρχών. θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ανοιχτή η αναφορά, να γράψουμε στις εθνικές αρχές, να ρωτήσουμε γιατί έλαβαν τη συγκεκριμένη απόφαση και όχι κάποιαν άλλη. Έγινε η μεταρρύθμιση, η μεταρρύθμιση αυτή πρόβλεπε και 200 σελίδες εξαιρέσεις. Γιατί δεν εκμεταλλεύτηκαν το περιθώριο που τους προσέφεραν αυτές τις εξαιρέσεις, για μένα είναι άγνωστο. Πρόταση λοιπόν, περισσότερη ενημέρωση. Ε, λυπούμε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει προσέλθει. Θα μπορούσε να ε, ρίξει κάποιο φως με την παρέμβασή της στην υπόθεση αυτή. Σας ευχαριστώ Πέτερ, ο κύριος Κόρχη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν είμαι μέλος της Επιτροπής Αναφορών, είμαι όμως Ιρλανδός Ευρωβουλευτής και συμμετέχω στην Επιτροπή Γεωργίας. Καλώς ήρθατε, λέει ο κ. Γιάρ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την πρότασή σας, κύριε Γιάρ, να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά του αναφερομένου και να γράψετε στο Ιρλανδικό Υπουργείο. Και προτείνω επίσης η αναφορά να διαβιβαστεί και στην Επιτροπή Γεωργίας και να ζητηθεί επισήμως γνωμοδότηση, διότι ως Ιρλανδός Ευρωβουλευτής ομολογώ ότι ντρέπομαι για το ότι ο αναφερόμενος χρειάστηκε να προσφύγει εδώ σε εσά, στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το θέμα του θα έπρεπε να είχε επιληθεί στο εθνικό επίπεδο. Μάλιστα, εδώ εξαντλώ τον κατάλογο εγγεγραμμένων αγορητών. Επανέρχομαι, θα επανέλθουμε μάλλον στην προηγούμενη σύντομα αναφορά δηλαδή το Ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας δεν έχει ακόμη απαντήσει στο αίτημα από την δική μας Επιτροπή Αναφορών. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες πληροφορίες, συντάσσουν απάντηση αυτή τη στιγμή, η οποία πρόκειται να μας έλθει σε λίγες ημέρες, ή πάντως σύντομα, σύντομα, ας το πούμε έτσι. Άρα, δεν θα χρειαστεί να ξαναγράψουμε στο Ιρλανδικό Υπουργείο ε, Γεωργίας, διότι είναι δουλειά την οποία κάνουν τώρα, απαντούν δηλαδή, υποτίθεται, συντάσσουν την απάντηση. Πάντως, η αναφορά έχει εξεταστεί α, στο κατάλληλο πλαίσιο στην Ιρλανδία. Αυτό που θα ήθελα να κάνω και απευθύνομαι και σε εσά, κύριε εκπρόσωπε του αναφερομένου, είναι να σας παρακαλέσω να εκφράσετε τη συμπάθειά μας, κατανόησή μας και ε, βαθύτατη συμπάθειά μας για τις ατυχίες στον αναφερόμενο. Βεβαίως ε, τηρούμε την αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου λάβουμε την απάντηση του Ιρλανδικού Υπουργείου Γεωργίας. Και βεβαίως αυτό που θα κάνουμε είναι να διαβιβάσουμε την αναφορά σας για ενημέρωση στην Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ε, ολοκληρώσουμε την συζήτηση της αναφοράς 1674. να επανέλθουμε τώρα στην αναφορά 1022 Σον Λόλες για την κακή εφαρμογή διατάξεων για την ενιαία καταβολή στα αγροκτήματα. Νομίζω ότι έχουμε επίσης ε, τους Κάνλον και Μέρφυ παρόντες. Έχετε το λόγο. Για πέντε λεπτά. Ευχαριστώ. Λέγομαι David Scanlon. Εκπροσωπώ τον Σον Λόλες. Σύντομο ιστορικό. 2010. Ο κύριος Λόλες είδε να μειώνεται κατά 90% η επιλεξιμότητα του αγροκτήματός του λόγω των ε, αγροτικών δραστηριοτήτων. Το 2012 αναφέρθηκε στην Επιτροπή Αναφορών η αναφορά του συζητήθηκε το 2014 και ζητήθηκε από τον Ιρλανδό Υπουργό Γεωργίας να προβεί σε ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη στο αγρόκτημα. Του είχε ζητηθεί να διεξαγάγει νοπή και ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Τον Ιανουάριο του 2015 το αρμόδιο γραφείο εξέτασε το αγρόκτημα, 250 περίπου εκτάρια, και κατέληξε στο ότι δεν είχαν καμία ένδειξη για να διαφωνήσουν με την ε, πραγματογνωμοσύνη του 2010 και ότι δεν υπήρχαν παρόντα ζώα στην ε, ημερομηνία της εξέτασης. Και διεξήγαγαν έρευνα για να δουν ποιες ήταν οι δραστηριότητες του 2010 και σημειώνουν επίσης ότι Λόλες και άλλοι μέτοχοι έχουν την υποχρέωση στη χειμερινή περίοδο να μην διατηρούν ζώα επί του αγροκτήματος αυτού. Τέσσερις ημέρες δηλαδή πριν από το γραφείο ε, ενστάσεων να κάνει την εξέταση, κάναμε εξέταση εμείς και εγώ και οι συνάδελφοί μου, εξετάζοντας ιδιαίτερα τις αγροτικές δραστηριότητες στο αγρόκτημα εκεί όπου το Agricultural Appeals Office δεν βρήκε ε, ενδείξεις αγροτικής δραστηριότητας, οι συνάδελφοί μου και εγώ ε, λάβαμε υπόψη τα περιτώματα των ζώων ως ένδειξη ε, αγροτικών δραστηριοτήτων. Στην διάρκεια της επίσκεψής μας βρήκαμε πολλά δείγματα περιτωμάτων και έχουμε μάλιστα καταγράψει και τις συγκεκριμένες συντεταγμένες τους με το σύστημα GPS. Χιλιάδες λοιπόν παραδείγματα ε, αγροτικής δραστηριότητας στο συγκεκριμένο αγρόκτημα. Επίσης η κατάσταση της χλώης εκεί δείχνει ότι ε, το αγρόκτημα έχει χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον για πολλά χρόνια. Έχουμε και φωτογραφικές αποδείξεις για πολλά χρόνια που αποδεικνύουν την ε, αγροτική δραστηριότητα στην τοποθεσία αυτή υπάρχουν, ε, υπάρχει ένας αριθμός εσφαλμένων παρατηρήσεων που έχει κάνει το ε, Υπουργείο Γεωργίας στην αρχική του έρευνα, τις οποίες έκανε και το Appeals Board, δηλαδή για την ε, αποκομιδή τύρφης, ότι δεν υπάρχουν εμπορικού χαρακτήρα, ότι δεν υπάρχουν δηλαδή εγκαταστάσεις για τα ζώα το οποίο και αυτό θεωρούμε ότι είναι εσφαλμένο. Είπαν επίσης ότι τμήματα του αγροκτήματος περιλαμβάνουν και τοποθεσίες όπου έχει ανέλθει το επίπεδο του έλους. Αυτό όμως θεωρείται μη επίπεδο. Δεν υπάρχει τέτοιου είδους τοποθεσία στο συγκεκριμένο αγρόκτημα. Άλλα λένε επίσης ότι μεγάλα τμήματα του αγροκτήματος είναι ακατάλληλα για ε, βόσκηση. Δεν υπάρχει όμως ποσοτικοποιημένος χάρτης για τις περιοχές αυτές και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχουν καν οι περιοχές αυτές. Τονίζω λοιπόν ότι, δεν υπά... Ε, ότι ε, έχει χαρακτηριστεί τοποθεσία ειδική προστασία σύμφωνα με το Natura 2010. Ένα θέμα το οποίο θέλω να θέσω ωστόσο είναι ότι υπάρχει πιθανότητα σύγχυσης, διότι η τοποθεσία αυτή αλλάζει πολύ από τους χειμερινούς στους θερινούς μήνες. Και όπως εξήγησα, ο κύριος Λόλες και οι άλλοι μέτοχοι δεν μπορούν να διατηρήσουν ζώα στην τοποθεσία αυτή στους χειμερινούς μήνες. Όμως δείτε εδώ στις εικόνες αριστερά χειμώνα, δεξιά ε, καλοκαίρι. Επιτρέψτε μου να δώσω το μικρόφωνο στην συνάδελφό μου Τρίσα Μέρφη, η οποία επίσης ε, εκπροσωπεί τον κύριο Λόλες και τους ε, συνεργάτες του. Ναι, πολύ σύντομα όμως γιατί μας τελειώνει ο χρόνος σιγά σιγά. Μάλιστα θα είμαι συντομοτάτη. Θα γνωρίζετε ότι η αναφορά είχε έρθει ενώπιον της Επιτροπής σας και ζητήθηκε να γίνει ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη, η οποία έγινε τον Ιανουάριο του 2014. Υπήρξε πρόβλημα ωστόσο με τη διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης με την έννοια ότι ο κ. Λόλες και δύο από τους αξιωματούχους που έκαναν την πραγματογνωμοσύνη συμμετείχαν και στην εξέταση πριν από την ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη. Δεν ήταν λοιπόν ανεξάρτητη πραγματογνωμοσύνη και αυτό ε, αφήνει σε δυσχερή θέση τον αναφερόμενο διότι τώρα δεν μπορεί να προσφύγει στο ανώτατο δικαστήριο ε, διότι τον εμποδίζουν οι διατάξεις του, της νομοθεσίας του 2001. Το Υπουργείο Γεωργίας προσέλαβε, ανέθεσε μάλλον στον ε, πρόεδρο του Συμβουλίου να προβεί σε πραγματογνωμοσύνη πριν από αυτήν που σας εξήγησα και τώρα αυτό προκαλεί παραπάνω δυσχέρειες στον ε, αναφερόμενο και για να γίνει ακόμα πιο δύσκολο το πράγμα για τον αναφερόμενο, το Ιρλανδικό Υπουργείο Γεωργίας έχει δώσει εντολή στον αναφερόμενο να προσφύγει στο Ιρλανδικό σύστημα δικαιοσύνης. Η δυσκολία για τον αναφερόμενο είναι ότι το Υπουργείο ε, Γεωργίας ανέθεσε στον επικεφαλής του Συμβουλίου να διεξαγάγει την πραγματογνωμοσύνη. Και αυτό εμποδίζει τον αναφερόμενο να προσφύγει για θέμα ε, νομικό στο ανώτατο Ιρλανδικό Δικαστήριο. Και μάλιστα η αναφορά έχει ήδη υποβληθεί στην Επιτροπή Αναφορών. Είναι δύσκολο λοιπόν να υποβληθεί νέα προσφυγή χωρίς τη συμμετοχή αξιωματούχων οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε προηγούμενες έρευνες. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Τώρα θέλουμε όλοι να ακούσουμε βέβαια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό, λέει η πρόεδρος Βίκστρομ. Ο κ. Κλίσον είναι παρόν. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, έχουμε από την μία πλευρά τον κύριο Σον ε, Ολέσε, ο οποίος είναι δικαιούχος ε, ενισχύσεων στα πλαίσια ε, της ΚΑΠ και από την άλλη πλευρά τους υπευθύνους υπεθεωρήσεων του Υπουργείου Γεωργίας, Επισητισμού και Θαλάσσης. Το σημείο εδώ αφορά την επιλεξιμότητα των γεών και κατά πόσον οι επιφάνειες που είχε δηλώσει ο κύριος Όλες έτσι ώστε ε, να ενταχθεί στο σύστημα ενισέας, ενιαίας ενίσχυσης Single Farm Scheme ή Single Payment εάν λέω το σύνολο των επιφανειών που είχαν δηλωθεί είναι επιλέξιμες. Ε, το πλαίσιο το νομικό ήταν ε, ο κανονισμός 73 του 99 που προέβλεπε ότι ένα επιλέξιμο εκτάριο ήταν οποιαδήποτε γεωργική επιφάνεια ε, που χρησιμοποιείται για λόγους γεωργικής δραστηριότητας ή σε περίπτωση ε, που χρησιμοποιούνται και για άλλες ε, δραστηριότητες θα έπρεπε οι κύριες δραστηριότητες να είναι γεωργικές. Όταν δεν εννοούμε με, την, με τον όρο γεωργική δραστηριότητα αναφέρουμε την κτηνοτροφία ε, ή ε, την γεωργία ή σε περίπτωση που δεν ε, χρησιμοποιούνται άμεσα για γεωργική παραγωγή έπρεπε αυτές οι επιφάνειες να διατηρούνται σε καλή γεωργική κατάσταση. τώρα, το ποιες ε, η απόφαση για την επιλεξιμότητα των γεών αφορά ε, τις εθνικές αρχές, κυρίως δε τους οργανισμούς που έχουν την δικαιοδοσία να χειρίζονται τις, ε, τις αιτήσει και να προχωρούν στις πληρωμές. Για να κάνουν κάτι τέτοιο οργανώνουν επιθεωρήσεις επιτόπου. Μετά από το τέλος αυτών των επιτόπου επιθεωρήσεων το 2010 λοιπόν το Υπουργείο Γεωργίας της Ιρλανδίας καθόρισε για την περίπτωση του κυρίου Λόλες το ποσοστό επιλεξιμότητας των γεών του. Σε αυτό το σύστημα, το οποίο είναι ε, κοινό σύστημα διαχείρισης, ο ρόλος των διαφόρων θεσμών ε, είναι σαφώς καθορισμένος η Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο καθορίζουν το γενικό νομικό πλαίσιο και επιθεωρούν κατά κάποιο τρόπο, με γενικό τρόπο τα κράτη-μέλη αλλά ε, η διαχείριση των φακέλων γίνεται σε καθαρά εθνικό επίπεδο. Οι εθνικές αρχές είναι αυτές ε, οι οποίες ε, θα πρέπει να λύσουν το ζήτημα και σε περίπτωση διαφωνίας τα εθνικά συστήματα εξοδικαστικού τρόπου επίλυσης διαφορών ή τα εθνικά δικαστήρια είναι υπεύθυνα για την επίλυση του ζητήματος. Δεν μπορούμε εδώ να πάρουμε θέση όσον αφορά το βασικό ζήτημα του του φακέλου αυτού που είναι η επιλεξιμότητα. Ο κύριος Τσόλος, νομίζω, Τσιόλος, ε, ο προηγούμενος ε, ε, επίτροπος υπεύθυνος για θέματα γεωργίας, νομίζω ότι είχε αναφερθεί ενώπιον της Επιτροπής σας το 2014 στο θέμα αυτό. Κατά αυτήν την έννοια λαμβάνομαι υπόψη τα νέα στοιχεία τα οποία έχει υποβάλει ο κύριος Λόλες, έτσι όπως κατατέθηκαν εδώ. Λαμβάνουμε επίσης γνώση του γεγονότος ότι αρχές 2015 η αρμόδια υπηρεσία υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας της Ιρλανδίας απήντησε στην Επιτροπή σας, αλλά παρόλα αυτά τα στοιχεία αυτά δεν, οδηγούν, δεν μας οδηγούν στο να αλλάξουμε θέση, δηλαδή ε, να ε, εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι τα ζητήματα αυτά είναι θέματα που εμπίπτουν στην εθνική αρμοδιότητα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος, για την ε, παρέμβασή σας. Εξακολουθώ πάντως εγώ να έχω πολλά ερωτηματικά. Τον λόγο έχει τώρα ο κύριος Κάρθη και νομίζω ότι ζητήσατε κι εσείς συνάδελφε τον λόγο. Και μετά κύριε Μακίνας. Ε, αυτή είναι... Πού ε, Κάπου, ψάχνοντας, τι να σου πω. Άντε, σε αφήνω να κοιτάξω το δικό μου, άμα θες. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ αναλυτικά ε, αναφέρθηκαν τα στοιχεία αυτά και πρέπει να ε, θυμηθούμε ότι η Επιτροπή μας ασχολήθηκε στο παρελθόν ε, με τα θέματα αυτά τα οποία σχετίζονται με τις επιτόπου επιθεωρήσεις Ακούσαμε και ε, τους δύο κυρίους που μίλησαν εξ ονόματος του αναφερομένου ε, και καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ορισμένα στοιχεία της αρχικής αποφάσεως δεν ήταν ε, σωστά. υπευλήθη η σχετική έφεση όσον αφορά την αρχική απόφαση στο αρμόδιο σώμα ε, αλλά ε, υπήρξε το πρόσκομα της ε, ανάμιξης ανθρώπων που είχαν ασχοληθεί ήδη προηγουμένως με το ζήτημα, πράγμα που δεν επιτρέπει στον αναφερόμενο να προσφύγει άμεσα στις εθνικές αρχές. Αλλά στην ουσία εδώ μιλάμε για ευρωπαϊκά χρήματα, για ευρωπαϊκούς πόρους και κατά την άποψή μου λοιπόν, ε, κατά αυτή την έννοια και αυτή η περίπτωση και άλλες παρόμοιες ε, αφορούν ή επιδρούν κατά κάποιο τρόπο στην αξιοπιστία εν τέλει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά και στην ε, προστασία της εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά ε, τις αποφάσεις ε, περιγεωργικών θεμάτων που θα πρέπει να βασίζονται σε ανεξάρτητη και αμερόληπτη βάση. Γι' αυτό λοιπόν ε, έπρεπε να είχαμε κάνει ε, μια αποστολή στην Ιρλανδία όπως το είχα ζητήσει αλλά δεν κατέστη δυνατόν. Τουλάχιστον όμως ε, θεωρώ ότι θα πρέπει να επανυποβληθεί το ερώτημα και επίσης ζητώ, για επίσκεψη δηλαδή επιτόπου στην Ιρλανδία και θεωρώ επίσης ότι θα πρέπει το ζήτημα αυτό να παραμείνει ανοιχτό και να διαβιβαστεί και στην Επιτροπή Γεωργίας έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση, ενδεχομένως μάλιστα και στην Ολομέλεια. Ε, ζητώ λοιπόν το αίτημα του αναφερομένου ε, να παραμείνει ανοιχτό, ε, να ξαναστείλουμε επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας της Ιρλανδίας ε, ε, σχετικά με το θέμα που μας απασχολεί σήμερα και οπωσδήποτε να συνεχίσουμε να ασχολούμεθα με το ζήτημα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. κυρία Μαγκίνες. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ξαφνικά γέμισε Ιρλανδούς αυτή η Επιτροπή. Είναι και αυτή την εβδομάδα η, η η γιορτή του Αγίου Πατρικίου, προστάτη της Ιρλανδίας, γι' αυτό. Κοιτάξτε τώρα, να πω πρώτα ποια είναι τα συμπεράσματά μου και μετά θα προχωρήσω στην ουσία. Πρέπει να πούμε και κάτι παραπάνω. Δεν αρκεί να στείλουμε επιστολή και να ζητήσουμε και άλλη προσφυγή, διότι νομίζω ότι σωστά τα είπαν οι ε, νομικοί σύμβουλοι. Εγώ νομίζω ότι χρειάζεται έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση και τον χειρισμό της, αλλά και για τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι επιθεωρητές που διεξήγαγαν την έρευνα, διότι φαίνεται να υπάρχει κάποια έλλειψη πίστης στη διαδικασία και στους υπαλλήλους που διεξήγαγαν την εξέταση. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε πώς έγιναν τα πράγματα αυτά. Να γράψουμε λοιπόν στις γεωρικέ αρχές, τον Υπουργό δηλαδή τον ίδιο, και να ζητήσουμε όχι απλώς επανεξέταση της υπόθεσης, αλλά και του χειρισμού της υπόθεσης, διότι αυτή η υπόθεση διαρκεί εδώ και χρόνια και οι αναφερόμενοι έχουν κολλήσει και δεν μπορούν ούτε πληροφορίες να βρουν. Η αναφορά λοιπόν να διατηρηθεί ανοιχτή. Θυμίζω και την αναφορά, την προηγούμενη αναφορά του ε, κυρίου Μακιού και η Κομισιόν Ενδεχομένω, Κοιτάξτε, δέχομαι ότι πρόκειται όντως για αρμοδιότητα της χώρας μέλους και το θέμα τίθεται μεταξύ αναφερομένου και χώρας μέλους. Όμως και η Κομισιόν έχει κάποια ε, υπόθεση εδώ, διότι αν υπάρχουν δυσκολίες για την χρήση των κριτηρίων επιλεξιμότητας και μεταξύ χώρων μελών αλλά και μεταξύ αγροκτημάτων, τότε πρέπει να εξετάσει το θέμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να γίνει αυτό για την ώρα και να ρωτήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν γνωρίζει ότι υπάρχουν και άλλες σχετικές υποθέσεις επιλεξιμότητα δηλαδή γεωργικών εδαφών παρόμοιες με την υπόθεση που έχουμε μπροστά μας. Είναι και ζήτημα και νομίζω της Ιρλανδικής Βουλής και της Αγροτικής της Επιτροπής. Και γιατί άραγε δεν επελήφθη μέχρι τώρα διότι θα έπρεπε να είχε τεθεί το θέμα και στο επίπεδο αυτό. Αντί δηλαδή να πούμε μόνον ότι, καλά, δεχόμαστε την άποψη τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτό δεν είναι δική μα αρμοδιότητα, α τα βρουν οι Ιρλανδοί μεταξύ του. Να διατηρήσουμε ανοιχτή την αναφορά, να ζητήσουμε από τι Ιρλανδικέ αρχέ να επανέλθουν, να επανεξετάσουν τη θέση του, αλλά να επανεξετάσει και η Κομισιόν την θέση τη. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα τουλάχιστον που ήθελα να θέσω υπόψη σα. Είναι πράγματι, λέει η Πρόεδρος, πολύ δύσκολη αναφορά. Πολύ δύσκολη και βεβαίως εξαιρετικά ευαίσθητη. Ο κύριος Φλάναγκαν και μετά να οροπληρώσουμε. Θα βάλω ένα όριο τώρα, διότι κλείνω τώρα τον κατάλογο των αγορητών και θα επανέλθω μετά στον αναφερόμενο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω. Λυπούμε που άργησα γνωρίζω την υπόθεση αυτή, έχω έρθει και σε επαφή με τους αναφερόμενους. Δύο πράγματα ε, εδώ. Αφενός, το Υπουργείο δεν φαίνεται να αμφισβητεί το γεγονός ότι η επιθεώρηση δεν ήταν και πολύ ανεξάρτητη. Και αν η επιθεώρηση δεν ήταν ανεξάρτητη και φαίνεται πως δεν ήταν ανεξάρτητη, φαίνεται Ούτως ή άλλως το φαίνεται, δεν είναι ωραία γιατί όπως είπε και ο ευρωβουλευτή Κάρκη πρέπει και να φαίνεται ανεξάρτητη. Αλλά εφόσον ε, δεν είναι ανεξάρτητη η Κομισιόν θα πρέπει να έχει κάποιο πρόβλημα σχετικά. Πάντω πρόκειται για γενικότερο θέμα όπως ε, το θέμα της επιλεξιμότητας των εδαφών είναι μέγα θέμα. Και να πει ότι η Κομισιόν δηλαδή ότι δεν έχει αρμοδιότητα επ' αυτού ή να δω μια στιγμή ακριβώς πώς λέει, να πει δηλαδή ότι δεν είναι δική της υπόθεση. Εγώ συναντήθηκα με αγρότες για θέματα επιλεξιμότητας και διόλου ξεκαθαρό δεν ήταν ποιος αποφασίζει. Δεν μπορεί να είναι μόνο το Υπουργείο, διότι αν το Υπουργείο κάνει κάτι, πώς να πω, παράνομο, φαντάζομαι ότι θα πάτε και θα τους πείτε ότι μπορεί να κάνετε τέτοια πράγματα. Άρα έχετε λόγο σε αυτό Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και άκουσα τι είπαν τότε στο Υπουργείο για την επιλεξιμότητα των εδαφών. Και αυτά που λέει και ο Μακάρκη δηλαδή, το θέμα αυτό ε, νομίζω ότι πρέπει να τεθεί υπόψη της Επιτροπής Γεωργίας και να εξεταστεί το θέμα αυτό ειδικά αλλά και πώς επαναλαμβάνεται σε άλλες περιοχές και να αντιμετωπιστεί συνολικά. Διότι είναι σαν να σου λένε οι γονείς σου πρέπει να πας στο κρεβάτι σου, αλλά δεν σου λένε πότε και αν δεν πας στη σωστή χρονική στιγμή, παρόλο που δεν σου έχουν πει πότε, σε μαλώνουν. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Πρέπει να γίνουμε σαφείς και συγκεκριμένοι γιατί διαφορετικά θα κάνουν οι αρχές ό,τι θέλουν, αλλά δεν είναι δυνατόν κάτι τέτοιο. Εδώ δεν είναι μόνο θέμα επιλεξιμότητας, είναι πολύ πιο γενικό. Ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπετε, δυστυχώς δεν έχουμε καθόλου χρόνο και έχουμε άλλη μια ισπανική αναφορά, την οποία αναλάξαμε. Προτείνω το εξής φαίνεται ότι όλοι οι συνάδελφοι συνάδουν στο και συμφωνούν στο να ε, κρατήσουμε ανοιχτή αυτήν την ε, αναφορά. Ε, θα πρέπει, γιατί σχετίζεται με την ίδια τη λειτουργία της ΚΑΠ. ωστόσο, οι υπεύθυνοι για την εκτέλεση της ΚΑΠ, κυρίως δε ε, όσον αφορά τις επιλεξιμότητες και την ενιαία ενίσχυση, είναι οι εθνικές αρχές θα πρέπει, θα πρέπει να ε, γίνει έφεση σε εθνικό δικαστήριο κατά της τελευταίας απόφασης. Αυτό πρέπει να κάνει ο ε, αναφερόμενος γιατί μόνο οι εθνικές αρχές μπορούν ε, να αμφισβητήσουν την ομιμότητα τέτοιου είδους απόφασης. Κύριε Φλάναγκαν, η Επιτροπή Γεωργίας έδωσε την άποψή της, τη γνωμοδότησε για το θέμα αυτό το 2010. 13 ήδη. Επομένως φαντάζομαι ότι μια και δεν άλλαξε τίποτα επί της ουσίας, εάν γνωμοδοτήσει πάλι τα ίδια πράγματα θα μας πει. Η Επιτροπή απήντησε, οι ε, αρμόδιες εθνικές αρχές έστειλαν ενδελεχέστατη απάντηση το Δεκέμβριο του 2015. Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι ναι, να κρατήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή, να επανέλθουμε προς την μόνιμη αντιπροσωπεία και να ε, ε, ξεκινήσουμε έναν ε, νέο διάλογο μαζί τους, να δούμε μήπως έχουν κάποια πρόταση να μας κάνουν. Αλλά να μην λησμονούμε ότι εμείς δεν είμαστε δικαστήριο και επομένως δεν μπορούμε <clears throat> περισσότερο, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε το θέμα αυτό παραπέρα. και μάλιστα θεωρώ ότι αν στείλουμε ξανά επιστολή στο, Υπουργείο, στο Εθνικό Υπουργείο της Ιρλανδίας ε, ε, που ασχολείται με τα θέματα γεωργίας θα είναι σχεδόν παρέμβαση στα εσωτερικά τους. Δεν μπορούμε εμείς να αμφισβητήσουμε αποφάσεις εθνικών αρχών ή αποφάσεις εθνικών ε, δικαστηρίων. Αλλά μπορούμε να στείλουμε όντως μία επιστολή ε, στην ε, Ιρλανδική μόνιμη αντιπροσωπεία εδώ στις Βρυξέλλες γιατί η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη. Ναι, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε να γίνει ε, νέα έρευνα, δηλαδή να τους ενθαρρύνουμε να γίνει νέα έρευνα με ανεξάρτητα άτομα αυτή τη φορά. Ναι, ναι, λέει η Πρόεδρος, οπωσδήποτε αυτό μπορούμε εντόνως να το υπογραμμίσουμε. Αλλά πραγματικά εδώ είμαστε στριμωγμένοι, δεν έχουμε πολύ περιθώριο, μεγάλο περιθώριο ελιγμών, γιατί εδώ μιλάμε για καθαρή αρμοδιότητα των εθνικών αρχών. Επομένως, με μεγάλη ταπεινοφροσύνη και με μεγάλη προ προσοχή και σύνεση μπορούμε να απευθυνθούμε σε αυτούς ε, παρακαλώντας τους, ζητώντας τους να ασχοληθούν με το θέμα αυτό. Δεν μπορώ να ξαναρχίσω την συζήτηση κύριε Φλάναγκαν. Έχουμε όπως σας είπα και προηγουμένως ακόμα μία αναφορά την οποία θα πρέπει να μελετήσουμε πριν ε, ε, λήξει η συνεδρίασή μας. Ε, επιστρέφουμε λοιπόν στο σημείο 10 της ημερησίας διατάξεως σχετικά με παρέμβαση Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την ρήπανση του ποταμού Γκαλέγο στην Αραγόνη. Στην Ισπανία. Θα δώσω το λόγο στον αναφερόμενο, <coughs> μια και επί της ουσίας έχουμε ήδη συζητήσει το θέμα της ρήπανση σε ένα άλλο σημείο της χώρας σας, αλλά παρόλα αυτά η ουσία παραμένει ίδια. Παρακαλώ λοιπόν να, να είστε σύντομος κύριε Σάντσες. Sí, gracias. Buenas tardes. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Αρχίζοντας θα ήθελα να δώσω δύο λεπτομέρειες σημαντικές για το λενδάνιο. Μιλούμε για ένα οργανικό συστατικό το οποίο παραμένει για πάρα πολύ μεγάλο χρόνο στην γη, στο νερό που θεωρείται και από την ε, Διεθνή Οργάνωση Υγείας καρκινογόνο και συμπεριλαμβάνεται στις πολύ μολυσματικές ουσίες. Εδώ έχετε την περιοχή του Σαβινιάνιγκο που υπάρχει το πρόβλημα. Έχετε έναν ε, ταμιευτήριο στον οποίο φτάνουν τα νερά τα οποία φτάνουν μέχρι το δέλτα του Εύρου. Πρέπει να πάει ίσως κάποια αποστολή για να δει πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Εδώ έχετε την περιοχή στην οποία ο ποταμός Γαλιέγο ε, χύνεται στον Εύρο στην περιοχή της ε, Σαραγώσα μικρές πόλεις που αφορώνται και επηρεάζονται είναι διάφορες. Πρώτα απ' όλα η Σαβινιάνιγκο, το εργοστάσιο στο οποίο, από το οποίο ξεκίνησε το πρόβλημα. Βλέπετε την πόλη μας και τα βουνά. Εδώ είναι το εργοστάσιο, το ένοχο, έτσι όπως είναι σήμερα. Δούλεψε από το 75 στο 89 η ημερομηνία για την οποία απαγορεύτηκε η χρησιμοποίηση του λινδανίου, αλλά συνέχισε τι δραστηριότητε του εργοστάσιο αυτό το 94. Από τότε μέχρι σήμερα, 22 χρόνια μετά δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο εγκαταλελειμμένο βρίσκεται στην μορφή που βλέπετε εδώ στο βίντεο. Έτσι είναι αυτό το ερείπιο. Σε αυτό το εργοστάσιο και στο οικόπεδο που το περιχλείτε μπορείτε να δείτε ε, κάποια ε, συστατικά από τα προϊόντα που κατασκεύαζε. Εδώ λοιπόν και 22 χρόνια έχουν αποθηκευτεί αυτά τα υλικά εδώ πέρα τα οποία ρηπαίνουν και βλέπετε πώς έχει η κατάσταση και πώς γίνεται η ρήπανση, η μόλυνση από αυτά τα κατάλοιπα. Άλλες εικόνες, 22 χρόνια μετά. Περί τίνος πρόκειται. Μιλούμε για απόβλητα ε, λινδανίου και στην περιοχή Μπαϊλίν, σε μια χωματερία έχουμε 150.000 τόνους, το Σαρδάς 140, 100 τόνους ε, στο ίδιο το εργοστάσιο και έρχεται και ένα, ε, μια περιοχή απορροής στην οποία έχουν συγκεντρωθεί όλα αυτά τα ποσά τελευταία χρόνια. Εδώ έχετε τους πολίτες που ζητούν τα δικαιώματά τους. Και γιατί ξαναρχόμαστε ακόμη μια φορά εδώ πέρα. Διότι απεδείχθη ότι είναι από τεχνικής και οικονομικής πλευράς ε, ανίκανες να λύσουν το πρόβλημα οι τοπικές μας διοικήσεις. Ζητούμε να μας προστατεύσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε κάθε πολίτης να μπορεί να έχει καθαρό πόσιμο νερό σε όλη τη ζωή. Και βεβαίως πρόκειται για ένα από τα βασικά και αναπαλωτρία τα δικαιώματα του κάθε ανθρώπου αυτό που ζητούμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θέλουμε δέσμευση. Δεύτερον, θέλουμε να σας καλέσουμε να επισκεφτείτε τις περιοχές αυτές ώστε να διτοποιήσετε πλήρως το πρόβλημα. Σας ζητούμε να λάβετε αποφάσεις. Σας ζητούμε βοήθεια οικονομική, ευρωπαϊκά κονδύλια για να μας βοηθήσετε να επιλύσουμε το πρόβλημα αυτό καθώς και το πρόβλημα των ε, ε, εκτάσεων που έχουν, των χερσαίων εκτάσεων που έχουν μολυνθεί, δεδομένου ότι υπάρχουν εκατομμύρια τόνοι γης που έχουν μολυνθεί. Αυτό ζητούμε από εσά, αυτό θέλουμε εξ όλων των συμπολιτών μας και για την προστασία του περιβάλλοντος και υπέρ του δικαιώματος του καθενός να έχει ποιοτικό πόσιμο είδωρ, αυτό ερχόμαστε να σας ζητήσουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή έχει το λόγο. Παρακαλώ να είστε πάρα πολύ σύντομος, διότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τα χρονικά μας όρια για σήμερα. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Και να αναφερθώ στην τελευταία γραπτή κοινοποίησή μας σε σχέση με την αναφορά αυτή. Όπως είπε και ο συνάδελφος προηγουμένως, σε σχέση με την αναφορά της ταμιευτήρα του Ογιόλα συμμερίζεται η Επιτροπή την ανησυχία που έχει προκληθεί από το πρόβλημα της μόλυνσης από το Λενδάνιο καθώς και στην περιοχή εδώ του ποταμού Γαλιέγο. Θα πρέπει παρόλα αυτά να ε, περιοριστούμε στα όρια των αρμοδιοτήτων που μας δίδει η κοινοτική νομοθεσία σε αυτή την περίπτωση και να πούμε ότι η οδηγία πλαίσιο απαιτεί σε τακτά διαστήματα να κάνουμε μετρήσεις τα ύδατα τα οποία υποψιαζόμαστε ότι έχουν μολυνθεί από το λινδάνιο, δεδομένου ότι όπως είπε και ο αναφέρον πρόκειται για μια πάρα πολύ επικίνδυνη ε, ουσία. Και θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μπορέσει να επανέλθει η καλή ποιότητα του πόσιμου είδου Το υδρολογικό πλάνο της περιοχής ε, του Εύρω προβλέπει διάφορες μετρήσεις ε, έτσι όπως το απαιτεί και η οδηγία πλαίσιο για την καθαρότητα του ύδατος και όσον αφορά τα μέτρα το 2015 η κυβέρνηση της Αραγών και της Ισπανίας ε, υπέγραψαν ένα σχέδιο βάση πρωτοκόλου δράσεων που θα ληφθούν για να είναι εγγυημένη ποιότητα. Και πιστεύουμε ότι έχουν εντοπίσει το πρόβλημα οι αρχές και ενεργούν. Η επικαιροποίηση του υδρολογικού ε, ε, σχεδίου του της του Εύρου θα φτάσει στην Επιτροπή μέχρι τα τέλη Μαρτίου και έτσι θα έχουμε την δυνατότητα να αξιολογήσουμε την πρόοδο που έχει επιτευχθεί για το θέμα αυτό που σας απασχολεί. Εξαιρετικά. Πολύ καλά νέα νέες πληροφορίες που δεν ήξερα. Εξαιρετικά τώρα το λόγο έχει η κυρία Αλβιόλ και μετά ο κύριος Σεβαστιά. κυρία Αλβιόλ. Ευχαριστώ. Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε ένα σαφές πρόβλημα ρήπανσης και κινδύνου για τη δημόσια υγεία και θα πρέπει να πούμε ότι οι δράσεις εκ μέρους των αρχών δεν επέλυσαν το πρόβλημα δεδομένου ότι συνεχίζεται να ανοιχνεύεται λινδάνιο στο νερό. Καμία από τις δράσεις που ανελήφθησαν δεν οδήγησε σε επίλυση του προβλήματος και, αδεμάς, ε, και εξάλλου στην περίπτωση του ποταμού Γαλλιέγου μεταφέρεται η ρηπογόνο ουσία. Πιστεύω ότι πρόκειται λοιπόν μια εξαιρετική δουλειά την οποία θα πρέπει να αναλάβουμε εμείς. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές οδηγίες που θα μπορούσαν ε, να βοηθήσουν, όπως η οδηγία πλαίσιο, η οδηγία που αναφέρει τις τεχνικές προδιαγραφές για την χημική ανάλυση και την παρακολούθηση της ποιότητας του νερού ε, τα θέματα της πρόληψης και της εμπορίας ε, προϊόντων που, που αφορούν την γεωργία. Πιστεύω ότι όπως και στην προηγούμενη περίπτωση έχουμε ανάγκη από μία ε, ευρωπαϊκή μελέτη για την ε, ε, μόλυνση σε όλη την Ευρώπη από τη χρησιμοποίηση του λινδανίου. Δεν πρόκειται για μία-δύο μεμονωμένες περιπτώσεις, αλλά για όλη την Ευρώπη. Θα θέλαμε λοιπόν να υποστηρίξουμε το αίτημα που γίνεται να υπάρξει διερευνητική επίσκεψη κοινοβουλευτικών εκπροσώτων στην περίπτωση του Ογιόλα Μπαρακάλδο καθώς και στην Αραγωνία στην περιοχή του ποταμού Γαλιέγο. Πιστεύω ότι καλό θα ήταν να οργανώσουμε μία αποστολή ώστε να επαληθεύσουμε επί τόπου περί τίνος πρόκειται και να συναντήσουμε τις αρχές ώστε να δούμε αν πραγματικά λήφθησαν οι απαραίτητε δράσεις. Πιστεύω επίσης ότι αυτό το οποίο μας ζητούν οι αναφέροντος είναι κονδύλια για να μπορέσει να καθαρίσει η περιοχή, διότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο αν δεν υπάρχουν οι καλτάλληλοι οικονομικοί πόλοι και ίσως η Επιτροπή Αναφοράς θα μπορούσε να υποδείξει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, αφιερώσει κάποια κοινοτικά κονδύλια για την απομόλυση. Και ξαφνικά βλέπω ότι η Επιτροπή μου από Ιρλανδική έγινε Ισπανική. Ο κύριος Σεβαστιά έχει το λόγο και μετά η κυρία Γιάλα Σάντερς. Παρακαλώ, συντομότατη, διότι είχαμε μια παρεμφερή αναφορά πριν από μια ώρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, θα προσπαθήσω και σε λίγο δεν θα έχουμε και διερμηνείς. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Πέρσι υπήρξε πρόβλημα μόλυνσης του ποταμού Γαλλιέγω και πάρα πολλά ε, χωριά χρειάστηκε να εφοδιαστούν με νερό το οποίο έφερναν ε, δεξαμενές. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόβλημα το οποίο είναι πραγματικό. Ακόμη δεν έχουν ανοιχτευτεί όλες οι δυνατότητες εστίασης στις ε, πηγές μόλυνσης έχουμε μεγάλες ποσότητες λινδανίου εκτός ελέγχου σε αυτή την περιοχή. Όπως στην προηγούμενη περίπτωση νομίζω ότι δικαιολογεί αυτά τα οποία ζητούν οι αναφέροντες. Δηλαδή ότι έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό ε, διαστάσεων πρόβλημα και δεν μπορεί καμία εθνική αρχή μόνη της να το αντιμετωπίσει αν δεν υπάρξουν ε, κοινοτικά κονδύλια για να λυθεί το πρόβλημα αυτό, το οποίο είναι γενικότερα και άλλες χώρες αφορώνται. Πιστεύω ότι μια ερευνητική επιτροπή και μια επίσκεψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτές τις δύο περιοχές θα μπορούσε να αποτελέσει την απαρχή ενός φιλόδοξου κοινοτικού προγράμματος ώστε να μην πολλαπλασιαστούν τέτοιου είδους περιπτώσεις. Γι' αυτό υποστηρίζουμε αυτά τα οποία ζητούν οι ατούντες και πιστεύω ότι μπορούμε να αναλάβουμε κάτι τέτοιο και να το υποστηρίξουμε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Γιάλα Σάντερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Και πάλι θα ήθελα να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα προηγουμένως. Μία ειδική ε, αναφορά και ένα αίτημα ειδικό η Επιτροπή ε, στις 22-23 ε, Μαρτίου θα πάρει το υδρολογικό σχέδιο το οποίο θα, τους, θα στείλει θα στείλουν οι αρμόδιες αρχές. Θα θέλαμε να το έχουμε και εδώ και θα θέλαμε να δούμε ποιες είναι οι νέες προτάσεις. Μας ενδιαφέρει αυτό και να επαναλάβουμε ότι μας ενδιαφέρει η αναφορά αυτή να αποσταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή Περιβάλλοντος να δει σφαιρικά όλες τις ε, πλευρές που άπτονται του θέμα αυτό Έχουμε να κάνουμε με ένα ευρωπαϊκό θέμα με αυτή τη μεγάλη μόλυνση. Και νομίζω ότι με μια τέτοια κρίση μπορεί να δημιουργήσουμε την ευκαιρία να λύσουμε γενικότερα το πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή αφορά και το θέμα αυτό και πλήγει την Ισπανία. Αλλά πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να ε, υποστηρίξουμε την υπόθεση αυτή ώστε να δούμε και να ανοιχνεύσουμε σε κάθε χώρα που υπάρχει σχετική μόλυνση πώς θα βοηθηθεί η κατάσταση. Χώρες σαν την Ισπανία δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν μόνε τους. Θα πρέπει λοιπόν να αποτελέσουν μέρος ενό ευρωπαϊκού σχεδίου δράση. Ε, το οποίο θα συνοδεύεται και από τα κατάλληλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Ευχαριστώ. Now to my vice... Εξαίρετα. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Αντιπρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ γρήγορα. Το θέμα αυτό μας απασχολεί εδώ και πολύ καιρό. Ε, και οι πληροφορίες που μας έδωσε το, η κεντρική κυβέρνηση, το Υπουργείο από το 2008 μέχρι το 2012 ε, είναι γνωστές, δηλαδή έχει υπάρξει ένα ε, συμβούλιο εμπειρογνωμόνων για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό, καθώς επίσης και ένα πρωτόκολλο συνεργασίας με την Αραγών, καθώς επίσης και μια συμφωνία για το 2015 17 εκατομμυρίων ευρώ ε, αυτό σημαίνει και γι' αυτό το λέω ότι δουλεύει ε, η Ισπανία ε, και παρότι, δεν, παρότι η Ισπανία από τον Ιανουάριο έχει υπηρεσιακή κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει αυτό που είπε η συνάδελφος Αγιάλα να αποσταλεί και αντιπροσωπεία της Επιτροπής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος ναι, είναι κάτι θετικό, θα το δούμε. Βέβαια για την ώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πάντως νομίζω ότι έχει ξεκινήσει μια καλή διαδικασία. Είναι λογικά τα όσα γίνονται. Και από εκεί και πέρα να δούμε τι θα πούν και οι συνάδελφοι της Επιτροπής Περιβάλλοντος και να αποφασίσουν. Thank you very much. And that concludes actually my... Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν έχω άλλον εγγεγραμμένο ε, αγορητή. Είναι παρόμοια με την αναφορά που μελετήσαμε προηγουμένως. Ε, προτείνω λοιπόν να προχωρήσουμε με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή να την αφήσουμε ανοιχτή και να δούμε ε, ποιο θα είναι το νέο υδρολογικό ε, σχέδιο το οποίο θα σταλεί στην Επιτροπή και τα λοιπά. Πέραν αυτού, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο εντομοκτόνο όπως το λινδάνιο, ίσως θα πρέπει να δούμε περισσότερο πόσο επικίνδυνο είναι. Γιατί προφανώς δεν υπάρχει μονάχα στην Ευρώπη, στην Ισπανία. Θα πρέπει να υπάρχει φαντάζομαι και στις υπόλοιπες 27 χώρες. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν των 28. Ίσως θα πρέπει να γίνει από το Policy Department ένα, μια μελέτη για το θέμα αυτό. Ίσως από με την Επιτροπή Περιβάλλοντος έτσι ώστε <coughs> να δούμε με ποιο τρόπο πρέπει να ε, προχωρήσουμε γιατί αυτό είναι ένα ε, πολύ σημαντικό ζήτημα για την ανθρώπινη υγεία και την υγεία εννοώ και στις 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τω μεταξύ όμως και μέχρι να έχουμε αυτήν την ε, ε, προτινόμενη ας πούμε έρευνα για το λιδάνιο στους 20, στις 28 χώρες ε, να προχωρήσουμε όπως σας είπα. Α, ναι, λέει η κυρία Γιάλα Σέντερ, ενδεχομένως να ενημερώσουμε σχετικά και την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ναι, ναι, ίσως για να είμαστε ισοδίκαιοι. Εν πάση περιπτώσει ό,τι γίνει πρέπει να γίνει ε, τώρα. Θέλετε κάτι να προσθέσετε. Ναι. Θα ήθελα να πω ε, να ε, ε, στείλουμε ξανά επιστολές στις αρχές οι οποίες δεν έχουν απαντήσει. Να τις στείλουμε ξανά και ενδεχομένως... We, know Can we mandate the secretary? Να τις επαναλάβουμε για να δούμε τι θα γίνει. Ναι, ναι, ναι, και θα αλλά είπαμε να περιμένουμε ε, πρώτα να έχουμε τα νέα στοιχεία, να στείλουμε επιστολές στη Ρέτζη και στην Έμβη. Και να έχουμε κατά νου ότι όταν θα έχουμε λίγο χρόνο και χώρο να ξεκινήσουμε μία πραγματική μελέτη για το θέμα αυτό. Έτσι να προχωρήσουμε. Συμφωνείτε? Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ και ειδικά, ειδικά θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διερμηνείς γιατί ήταν πολύ ε, ε υπομονετικοί μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.